Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε στις πληροφορίε. Είναι πια 9 η ώρα και ο χρονός μας πιέζει. Οπότε μπορούμε καταρχήν να κάνουμε την αξιολόγηση της χρήσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ο κύριος Χαΐς δεν θέλει να λάβει το λόγο παρόλο που είναι εισηγητής. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ε, με την ε, ψηφοφορία, γιατί στα αγγλικά θα γίνει για να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ξέρετε όλοι τι ψηφίζουμε. Είναι η γνωμοδότηση Hayes. Είναι η έκθεση Hayes. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Καταπίπτει. Τέσσερα σε δύο μέρη, πρώτο τμήμα υπέρ, δεύτερο, με κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, ηλεκτρονικά παρακαλώ, το δεύτερο τμήμα της 4. Έχουμε 11 ε, κάρτες που ψηφίζουν. Τι βλέπουμε εδώ, 9. Λοιπόν, έληξε. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Τροπολογία. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά αποχές. Παρακαλώ την 7 ηλεκτρονικά. 9, 10, 11, 12 κάρτες. Βελτιωνόμαστε. Έληξε. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, απορρίπτεται. Συγγνώμη, κάτι άλλο κοιτάγα. 6 υπέρ. Συγγνώμη, 8. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ και την 8 ηλεκτρονικά. Σας παρακαλώ πολύ. Τροπολογία 8 ηλεκτρονικά. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τη 14 παρακαλώ ηλεκτρονικά, γιατί έχουν αλλάξει τα νούμερα των ε, βουλευτών και αλλάζουν και οι θέσεις που κάθονται. Έληξε, εγκρίνεται. 15 και 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 20 υπέρ. Στο συμβαστική 2 παρακαλώ, ηλεκτρονική, ο ηλεκτρονικός έλεγχος, ψηφίζουμε. Πέρας, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ απορρίπτεται είναι ξεκάθαρο την 22η παρακαλώ έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ηλεκτρονικά ναι, μάλιστα απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την 24 λοιπόν ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Η 25 έχει Απερίφθη. Την 25 παρακαλώ. Επιστρέφουμε στην 25 και την ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Η 25 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 1. Δεν ψηφίζουμε. Ρέτζι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 για την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης άρχεται. Πέρας και εγκρίνεται. Ομόφωνα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία, την επόμενη. Τον τελωνιακό εξοπλισμό εισηγητή είναι ο κύριος ε, Άλλη. Γνωμοδότηση τη ΣΥΜΚΟ. Θέλει ο εισηγητή να λάβει το λόγο. Όχι. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Με το σημείο 11. Θέσπιση, όχι. είναι κομμάτι του ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, ε, θέσπιση το Μεσό Χρηματοδοτικής Στήριξης για τον Εξοπλισμό των Ολιακών Ελέγχων, κύριε Άλλη. Ε, μιλάμε για το σημείο 11 της ημερησίας διάταξης, ε, τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ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 Προφορική τροπολογία 1. Δεν υπάρχουν ενστάσεις υπέρ. Είστε κατά της προφορικής τροπολογίας. Είστε δεν είστε. Προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχουν ενστάσεις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 καταπίπτει. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά κατά αποχές ε, απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ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 Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 17. Πέρασε. Ελέγχου. Συγγνώμη, δεν το είδα. 18 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές. Ε, εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές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 αποσύρεται επί όλη της γνωμοδότηση με ονομαστική ψηφοφορία. Έρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορία 17 προς 1 ο κύριος Τάραν δίνει μια ψήφο υπέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 12 το σχέδιο γνωμοδότησης προς την ΙΜΚΟ για το Τολωνιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας. Συζητητής ο κύριος κλίντ θέλει τον λόγο. Όχι, ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ,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 κατά αποχές να το επαληθεύσουμε να επαληθεύσουμε το 28 Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ψηφίσει, τέλος. Και τα αντίστοιχα υπέρ, άρα εγκρίνεται. Ναι, ναι, εγώ καθορίζω τις εξελίξεις. Ναι, συμβαίνουν αυτά. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές να το ξαναδούμε το 30 πέρας και τάραντ κατά απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εσείς υπέρ μάλιστα εγκρίνεται εύκολο. Να το δούμε, να το ξαναδούμε. Ωραία. 31, να το επαληθεύσουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Να το δούμε και θα το επαληθεύσουμε. Όχι, νομίζω ότι απορρίπτεται. Ναι, ναι, απορρίπτεται και η γραμμοδότηση στο σύνολό της με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας 18 υπέρ μία ψήφος κατά συγχαρητήρια. Τελευταία ψηφοφορία είναι για την Άγκαρη. Ο κύριος Στεχόφσκι είναι ο εισηγητής. Θέλετε τον λόγο. Όχι. Μία μικρή ψηφοφορία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 σε 2 μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρο δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές να το απελθέψουμε εγκρίνεται Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η δρομοδότηση του σύνολό της με ψηφοφορία έρχεται και πέρασε 17 υπέρ, μία ψήφος κατά συγχαρητήρια στον εισηγητή τελείωσε η ψηφοφορία παρακαλώ διαλυθείτε ησύχως εάν δεν θέλετε να ακούσετε τον κύριο Επίτροπο Καλημέρα σας κύριε Επίτροπο. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Καλώς ήρθατε κύριε Επιτροπέ, χαιρόμαστε που είστε εδώ. Σημείο 14. Απαλλαγή της ε, Κομισιόν για τον προπολογισμό της έρευνας για το δικαστήριο κ. για το ελεγκτικό συνέδριο με συγχωρείτε. Ο κ. Χένιγκ Μάιερ θα το παρουσιάσει. Αλλιώς μπορούμε να... Κύριε Μάιρ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρέσλε, Πρόεδρε της Επιτροπής. Είμαι ο Άλεξ Πρένιν και είμαι μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του ελέγχου μας για το κεφάλαιο 5 ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για το 2017. Έχουμε προετοιμάσει κάποιες ε, διαφάνειες για να σας παρουσιάσουμε τα βασικά μας ευρήματα. Το πρώτο είναι ότι η συνολική δαπάνη για το κεφάλαιο αυτό είναι 21,4 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανέμεται στην έρευνα σε μεγάλο βαθμό το μεγαλύτερο κομμάτι είναι έρευνα 70% συγγνώμη και άλλοι τομεί είναι οι μεταφορές, ε, το διάστημα, λοιπές δράσεις, η εκπαίδευση με μικρότερα ποσοστά. Το μεγαλύτερο λοιπόν κομμάτι είναι η έρευνα. Κατά 53% συγγνώμη. Όπως είδαμε λοιπόν η έρευνα είναι 53%. Το δείγμα μας ήταν 130 συναλλαγές ε, που κατανέμονται σε 91 για έρευνα και 70% δηλαδή και 39 για τα λοιπά προγράμματα. Σε αυτό το τομέα πολιτικής Υπάρχουν διάφοροι δικαιούχοι, ε, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, δημόσιοι, κρατικοί φορεί, ε, ιδιωτικέ εταιρείε και μικρομεσαίες επιχειρήσει. Όπω επίση και αυτό είναι σημαντικό, φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είχαμε 18 ελέγχου σε κράτη-μέλη και 5 σε χώρε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε την εξέλιξη του συντελεστή σφάλματος για το κεφάλαιο 5, μπορούμε να παρατηρήσουμε καθοδική τάση. Παρατηρούμε συντελεστή σφάλματος για το 2017 της τάξης του 4,2%. Η διαφορά με τα τελευταία χρόνια στατιστικά δεν είναι σημαντική. Ο αριθμός των δειγμάτων που λάβαμε φέτος ήταν 130. Για το πλαίσιο τώρα αυτού του ελέγχου και του αποτελεσματός του, καλό είναι να δει κανείς την ευρύτερη εικόνα των πορισμάτων του ελεγκτικού συνεδρίου. Εδώ απεικονίζεται ο ελεγχός μας ε, σε συνοπτική μορφή. Μπορεί να δει κανείς ότι τα μηχανισμοί ε, επιστροφής κόστους ε, έχουν, είναι πιο επιρρεπείς σε σφάλματα Και αυτό αποτελεί σημαντική ε, διαφορά για το ελεγκτικό συνέδριο. Κάτι άλλο που παρατηρούμε είναι η αργή σταδιακή ε, λήξη του FP7 πρόγραμματος πλαισίου 7 Έχουν αυξηθεί οι δράσεις για το Horizon 2020 παρότι παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. 38 σε σχέση με τις 53 του προγράμματος πλαισίου 7 οπότε ακόμα ε, βλέπουμε το πρόγραμμα πλαίσιο να κατέχει σημαντικό κομμάτι και του χρόνου ο συνάδελφός μου ε, που θα αναλάβει θα δει τον αριθμό να αλλάζει σημαντικά υπέρ του οριζόντα 2020 και εκεί θα είναι πιο σαφές ε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από την απλούστευση του οριζόντα 2020. Uh, είναι σημαντικό να δούμε ότι είναι λίγο ανησυχητικά υψηλό ο συντελεστής φάλματος. Πάντα ελπίζει κανείς ότι θα μειωθεί σημαντικά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε προσδιορίσει τα οκτώ μεγαλύτερα σφάλματα που αντιστοιχούν ε, συντελεστή σφάλματος 2,5%. Όλα σχετίζονται με την έρευνα. Πέντε από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και τρία από τον οριζόντα 2026 ε, οφείλονται σε λάθος υπολογισμό του δαπανών προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι ο υπολογισμό ε, των δαπανών προσωπικού είναι περίπλοκος ε, και ε, εκεί μπορεί να παρουσιαστούν σημαντικά ασφάλματα. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι πέντε δικαιούχοι του δημόσιου τομέα σε αυτή την ομάδα των σφαλμάτων υψηλού κινδύνου και τρεις είναι οι δικαιούχοι από τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μία μη κερδοσκοπική οργάνωση. Πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι Μεγάλο ποσοστό δικαιούχων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατατασσόταν εντός των τομέων δαπανών υψηλού κινδύνου. Ε, ένα από την ε, Ελβετία, ένα από την Νορβηγία, ένα από την Τανζανία και ένα από τι ΗΠΑ δικαιούχοι. Δύο σφάλματα διαβιβάστηκαν ω υπόθεση στην Όλαφ, η οποία ελπίζουμε ότι θα ερευνήσει τις υποθέσεις αυτές. Συνοπτικά πρέπει να σημειωθεί ότι το, οι δαπάνες προσωπικού είναι η βασικότερη πηγή σφάλματος. Χρειάζεται λοιπόν βελτίωση ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό με φέρνει εν συντομία στις συστάσεις μας. Ε, η πρώτη μας σύσταση είναι να διευκρινίσουμε τους κανόνες και τις μεθοδολογίες ε, για το κόστος προσωπικού και ειδικότερα για ορισμένε χώρε, να ψάξουμε να βρούμε δηλαδή πού βρίσκονται τα προβλήματα, σε ποιε χώρε και πώ μπορούν να επιληθούν. Η σύσταση 2, βελτίωση του επίπεδου ευαισθητοποίησης μεταξύ δικαιούχων ε, των κανόνων επιλεξιμότητας, ειδικότερα κάνοντα μια σαφή διάκριση μεταξύ ενό συμβολέου υλοποίηση και ενό ε, δεύτερου συμβολέου, ε, σύσταση 3, υλοποίηση των συστάσεων IAS, περισσότερο τεχνική φύση αυτό. των διεθνών λογιστικών προτύπων. Δηλαδή, όπω βλέπετε, θα χρειάζονται προσπάθειε για να μειωθεί ο συντελεστή σφάλματο σε αυτόν τον τομέα πολιτική. Όπω ξέρετε, το ελεκτικό συνέδριο έχει κάνει δύο προσπάθειε να παράσχει ε, σημαντικέ πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο μέσω τη απλούστευση. Στην νομοθετική διαδικασία έχουμε παρερεύει με ένα ενημερωτικό έγγραφο για την απλούστευση το Μάρτιο του 2000, ε, στις 26 Μαρτίου φέτος. Και πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία έκθεση ελέγχου για τα μέτρα απλούστευσης. Οι εκθέσεις αυτές ε, εκπονήθηκαν σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν, ώστε να παρουσιάσουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες ε, για θέματα απλούστευσης. Ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα φέρει αποτέλεσμα στο μέλλον ε, με μείωση σημαντική του συντελεστή σφάλματος. Ήθελα απλά να σας δείξω τα παραρτήματα, δεν θα τα παρουσιάσω λεπτομερώς για τα συνόψεις, αλλά πιστεύω ότι λέει πολλά αν διαβάσει κανεί ε, αυτά τα παραδείγματα, καταλαβαίνει πολλά, αντιλαμβάνεται, αποκτά μια εικόνα του ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Πρόεδρε, είμαι πολύ ικανοποιημένο που σας παρουσιάζω αυτό το αποτέλεσμα και με μεγάλη μου χαρά θα απαντήσω στι ερωτήσεις σας. Σα ευχαριστώ για την εισαγωγή σας και την σαφήνειά σα. Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω εκτός από τον κύριο Επίτροπο και τον κύριο Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Πακέ. Κύριε Επίτροπο, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλερ ε, κυρία Σέντερ, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής και βεβαίως στο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ήθελα να πω τα εξή. Νομίζω πως είναι η τελευταία φορά που ο κ. Μπρένινγκ Μάιερ είναι ο υπεύθυνο για την έκθεση, για την καινοτομία και την έρευνα και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια για τις αιτήσεις εκθέσεις, για τις ειδικέ εκθέσεις, για την ε, καινοτομία και τα σχετικά ε, σεμινάρια, τα ελεγκτικά, πραγματικά φέρατε τη διαφορά και έχουμε βελτιώσει πολλά στοιχεία της δράσης μας γιατί μας πείσατε, γιατί μας ενθαρρύνατε και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για στο μελλοντικό σας ρόλο. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βρίσκομαι σήμερα για να συζητήσουμε την έκθεση τον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2017 και είμαι πεπισμένο για την σημασία που έχει για την Ευρώπη η έρευνα και η καινοτομία. Θα πρέπει την πρόκληση της προώθησης αυτής ε, και τη σωστή οικονομικής διαχείρισης των σχετικών ταμείων να τη θέσουμε ε, στον πυρήνα του προγράμματό μας. Και είχα έρθει ε, μέσα στη χρονιά για να σας πω πιο ανεπίσημα τις επιτυχίες που σημειώθηκαν φέτος και που αποδεικνύουν την πραγματικότητα και τον αντίκτυπο των όσων κάνουμε. Είμαστε πολύ περήφανοι που φέτος για μια χρονιά ακόμα στηρίξαμε ένα από τα βραβεία Νόμπελ. Ο Ζεγάρ Μογό είναι άτομο το οποίο εμείς έχουμε επιχορηγήσει. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και με τις ενισχύσεις αυτές μπόρεσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα λέιζερ και ο τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε για παράδειγμα ε, για ε, εγχειρήσεις ε, μοιοπίας ε, μείωπες όπως εγώ για παράδειγμα ή άνθρωποι που υποφέρουν από καταράκτη μπορούν να εγχειριστούν και άλλαξε τον τρόπο που γινόταν με αποτέλεσμα να του δοθεί το βραβείο Νόμπελ. Και ήταν καταπληκτικό το γεγονό ότι ήταν τα ευρωπαϊκά χρήματα που του επέτρεψαν να κάνει αυτή την έρευνα. Και αυτό δεν είναι το τελευταίο. Έχουμε πάρα πολλέ εφαρμογέ από την ε, πυρηνική σχάση ε, μέχρι νανοτεχνολογία σε υλικά με ολόκληρη γκάμα τεχνολογικών προϊόντων που είναι επιτυχία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσα στη χρονιά είχα την ε, τύχη να συναντήσω τον Σεντρίκ Λαμλάου που είναι εμπειρογνώμονας ερευνητή σε θέματα καρκίνων που εργάζεται στο Βέλγιο, στο Βέλγιο και ε, για τον καρκίνο φέτος σήμερα έκανε μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις γιατί ανακάλυψε ανακάλυψη περίπου δύο ειδικητάρων. Δηλαδή, ε, κύτταρα που αναπτύσσουν τον καρκίνο και κύτταρα μεταστατικά. Πάντοτε θεωρούσαμε πω είναι τελείω διαφορετικά αυτά τα κύτταρα και τώρα ο ίδιο κατάλαβε πω υπάρχει ένα μηχανισμό και μπορεί να είναι ένα κύτταρο το οποίο μπορεί να αλλάξει και από πρωτογενή καρκίνο να γίνει μεταστατικό. Γνωρίζοντα λοιπόν το μηχανισμό, μπορεί κανεί να διακόψει τη διαδικασία μετάσταση, ε, αλλάζοντα τα κύτταρα αυτά, ώστε να μην είναι πλέον μεταστατικά. Το ξέραμε αυτό και στο παρελθόν και ξέρατε πως αν ε, έχετε ένα μεταστατικό κύτταρο αυτό θα προκαλεί όλο και περισσότερες μεταστάσεις. Ε, αυτό λοιπόν είναι κάτι καταπληκτικό και είναι πάλι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το επέτρεψαν να κάνει αυτή την ανακάλυψη. Τέλος, από το Ινστιτούτο Max Planck ε, συνάντησα τον Peter Seaborg που έχει βρει ένα εμβόλιο για τους ανθρώπους που υποφέρουν από πνευμονία. Ε, πνευμονία ε, που προέρχεται από τον ε, βάκυλο του στρεπτόκοκου που σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει στη φάση την δοκιμή με ζώα στο εργαστήριο και σύντομα θα περάσει και στις δοκιμές με ανθρώπους. Με πειραματόζωα λοιπόν τώρα, με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτές είναι επιτυχημένες ιστορίες που έχουν να κάνουν και με ανθρώπους που είναι τελείως ε, ε, ε ξεκάθαρα επιστήμονες και με ανθρώπους οι οποίοι απλώς αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε για την ε, επιστήμη. Τώρα, για τη γυναίκα που πήρε το βραβείο για την καινοτομία στις γυναίκες το 2018. Έφτιαξε ένα ρομποτάκι, και αυτή είναι η άλλη περίπτωση που σας είπα, που βοηθάει τους ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι και βοηθάει τα παιδιά και τους ε, νέους ενηλικές που έχουν ε, μακροχρόνιες παθήσεις που θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουν και που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν και να δουν τους φίλους τους. Δεν μπορούν να κάνουν γυμναστική, δεν μπορούν να πάνε σχολείο, δεν μπορούν να περάσουν από εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ε, θεοδομένο για τους ίδιους δεν γίνεται. Και λόγω αυτού του ε, έργου που λέγεται καθόλου απομόνωση, ενώ isolation της Κάρολ Ντόνοβαν, τα παιδιά αυτά έχουν κάποιον με τον οποίο μπορούν να αποκτήσουν μια σχέση και να τους βοηθήσει, ε, για παράδειγμα, ε, μαθησιακά κτλ. Και αυτή τη στιγμή 650 παιδιά στην Ευρώπη το χρησιμοποιούν. Τέλος, πέρσι η Χριστίνα Ζεβανόβα από τη Βουλγαρία έφτιαξε ένα τάμπλετ για τους τυφλούς που επίση κέρδισαν ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Οπότε αυτέ οι ιστορίε εμεί θα πρέπει να τι επικοινωνούμε, είναι πολύ σημαντικέ και είναι πολύ σημαντικέ και για το μέλλον μα. Πριν από δύο περίπου εβδομάδε ξεκινήσαμε τη στρατηγική για τη βιοοικονομία και εγώ πρέπει να σα πω πήγα στη συνέντευξη τύπου στο κτίριο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορώντα ένα πράσινο φουλάρι που είναι εξίσου καλό με οποιοδήποτε άλλο φουλάρι αλλά δεν είναι ένα συνηθισμένο ύφασμα είναι φτιαγμένο από πούλπα ξύλου που μετατρέπεται σε ύφασμα. Πράγματα τα οποία εμείς αναπτύσσουμε στην Ευρώπη, έχουμε την ηγετική θέση, θα πρέπει να τη διατηρήσουμε και θα τα καταφέρουμε πιστεύω στο μέλλον. Οπότε, πριν μπούμε στα νούμερα, θα ήθελα αυτά τα παράδειγμα να τα ξέρετε για να ξέρετε τι είναι αυτό που αλλάζει τη ζωή μας. Κοιτώντας την έκθεση για τις δαπάνες του 17, και αν τα δείτε αντίστροφα θα δείτε πως ουσιαστικά ρίχνετε μια ματιά και ταινίζετε το μέλλον. Η πρόταση για το Horizon Europe ε, με τις συστάσεις της έκθεσης Λαμή είναι αυξάνουμε τις επενδύσεις στην έρευνα, ξεκάθαρο αυτό, οικοδομούμε μια πραγματική καινοτόμο πολιτική για να έχουμε νέες αγορές, παιδεία για το μέλλον και επενδύσεις στους ανθρώπους. Και βεβαίως μία προσέγγιση που θα βασίζεται σε μέτρηση αντικτύπου για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Επενδύσεις λοιπόν στην τεχνολογία και στην έρευνα και στην καινοτομία είναι η καλύτερη εναλλακτική για την Ευρώπη και το Horizon Europe στην πρόταση που υποβάλαμε είναι ένα απόσταγμα των εμπειριών μα και από τι δικέ μας έκθεσης αξιολόγηση και τι εκθέσει του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να τα πάμε καλύτερα για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μπρένιγκ Μάιερ που δημοσίευσε πιο σύντομα αυτή την έκθεση, ε, μάλλον το σημείωμα briefing, όπω επίση και την έκθεση για το Horizon 2020. Το έγγραφο briefing, το σημείωμα αυτό μα βοήθησε και μα βοήθησε να προετοιμάσουμε και τι νέε προτάσει για το Horizon Europe και η ίδια η έκθεση καταλήγει να φτάνει στα χέρια μας την κατάλληλη στιγμή για να προετοιμάσουμε μια πιο απλή και πιο αποτελεσματική στρατηγική εφαρμογής για το μέλλον. Κλείνει ως συμπέρασμα έκθεση λέγοντας πως η πλειοψηφία των μέτρων απλούστευσης που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η έκθεση λοιπόν συμπερασματικά καταλήγει και παραθέτω και λυπάμαι που βιάζομαι για τους γερμηνείς η πλειοψηφία των μέτρων απλούστες που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αποτελεσματικά στη μείωση του διοικητικού βάρους για τους δικαιούχους του Horizon 2020. Παρόλο που δεν ήταν όλες οι δράσεις αυτές που έδωσαν τα αποθητά αποτελέσματα και τις ευκαιρίες ε, έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω είναι δίκαιο το συμπέρασμα. Πετύχαμε αποτελεσματικά αποτελέσματα απλούστευσης. Οι επιδόσεις μας, το 81% των δικαιούχων το είπε το Ελληνικό Συνέδριο, θεωρούν πως είναι πιο απλό από ότι ε, το ε, πρόγραμμα πλαίσιο ε, το 7ο. Αλλά θα πρέπει να πάμε πιο πέρα, να λάβουμε υπόψη τα ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου, να δούμε τις νομοθετικές προτάσεις και θα το κάνουμε αυτό στη διαδικασία δραστηριοποίησης για την εφαρμογή του προγράμματος. Η έμφαση αυτή ε, για την αποδοσή και για τον αντίκτυπο δεν σημαίνει πως θα δώσουμε λιγότερη σημασία στα θέματα τα εφαρμοστικά. Και αυτό με οδηγεί στο ε, ποσοστό σφάλματος για τη χρονιά αυτή. Το ποσοστό σφάλματος για το κεφάλαιο ολόκληρο είναι στο 4,2% όπως μας είπε ο κ. Μπράνινγκ Μάγερ. Και αυτό είναι περίπου το ίδιο με την περασμένη χρονιά. Αλλά έχει μειωθεί και θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθα, το 14 να σας δω, έχει πέσει από το 5,6% το 2014. Και ελπίζω πως αυτή ε, η τάση θα συνεχιστεί. Το ποσοστό σφάλματος έχει να κάνει κυρίως με τις δαπάνες του προγράμματος πλαίσιο ε, του εβδόμου, γιατί βεβαίως ε, έχουν κάποιες δαπάνες από το Horizon 2020 το δείγμα, αλλά οι 53 πράξεις ήταν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και για το Horizon 2020 εμείς έχουμε κάνει ένα πρώτο υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος που θα βρείτε στην έκθεση ε, ε, δράσεων για το 2017. Και από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε, από το αντιπροσωπευτικό σφάλμα για το Horizon 2020 είναι πως είμαστε στο 2,8% και αυτό θα συγκριθεί με το 5,6% στο παρελθόν. Και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω πως αυτά είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις. Και οι αξιολογήσει μας είναι ακριβώς σε πολύ ε, πρώιμη φάση της δαπάνης για το Horizon 2020. Μπορεί αυτό να αλλάξει, να αντιστραφεί αυτή η τάση, αλλά οι ενδείξεις που έχουμε είναι πως η απλούστευση που εισήχθη είχε επίπτωση και το εναπομείνουν σφάλμα λαμβάνοντας υπόψη και τις ανακτήσεις και τα υπόλοιπα σφάλματα μας φέρνει στο 2,24% για το Horizon 2020. Και αυτό σε σύγκριση με το 3% για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και αυτό θα το βρείτε πως είναι στο χαμηλό σκέλος του στόχου που έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν παρουσίασε τις προσδοκίες για το Horizon 2020 που ήταν μεταξύ 2 και 5%. Να σχολιάσω τώρα ε, εντάχει και τα σχόλια ε, τα, της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καταρχήν, απλούστευση. Αναγνωρίζει το ελληνικό συνέδριο πω και η ετήσια έκθεση και οι ειδικέ εκθέσει για την απλούστευση για το 2020 είναι καλύτερε. Δηλαδή, χρηματοδότηση πιο απλή κανόνε σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Παρόλα αυτά, βρίσκει πολλά σφάλματα και θεωρεί πω οι κανόνε για τα ε, κόστη προσωπικού είναι δύσκολο και να κατανοηθούν και να εφαρμοστούν. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο, συμφωνούμε, και θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, και να περάσουμε στην εφαρμοστική φάση ε, του ε, Horizon 2020. Εκεί δημιουργήσαμε όλους τους κανόνες, διαδικασίες και συστήματα για να διαχειριστούμε τις επιχορηγήσεις για έρευνα και να περάσουμε στο στην ηλεκτρονική διαχείριση. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση που θα έχουμε ε, ένα καταποκοπή ποσό για τα έμεσα κόστη και με μία δόση αποπληρωμή όλων των δαπανών έρευνας. Είναι πιο απλό, είναι παντελώς ψηφιακό το σύστημα αυτό και κάνουμε ό,τι μπορούμε πιστεύω. Οπότε, στα πλαίσια του δεύτερου κύματος απλουστεύσεων, τα, ε, κόστη προσωπικού και αμοιβών προσεγγίζουμε το σύστημα, το λογιστικό που ακολουθούν οι όχι και ξεκινήσαμε με κάποια πειραματικά πιλωτικά σχέδια για καταποκοπήν ενίσχυση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, υποχρεώσει υποβολή εκθέσεων για το προσωπικό, έτσι ώστε και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και όσοι κάνουν καινοτομίε να μπορούν να μπρουν και στην χρηματοδότηση. Και γι' αυτό στη δοκιμαστική φάση έχουμε και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία. Η τάση είναι καλή. Δεύτερον, για να αποφεύγουμε τα σφάλματα. Το δικαστήριο λέει πως ο αριθμός, αριθμός σφαλμάτων θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί πριν τη πληρωμή λόγω αδυνομίας στα πιστοποιητικά ε, τα ελεγκτικά και γι' αυτό επειδή το αναγνωρίσουμε ξεκινήσαμε μια επιπλέον δράση επικοινωνίας και βεβαίως οι συστάσεις οι ελεγκτικές ενισχύονται και θα πρέπει και τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου να τις εφαρμόσουν οι δικές μου ελεγκτικές υπηρεσίες. Θα είμαστε σαφείς λοιπόν πως αυτά τα οικονομικά ασφάλματα ε, δεν είναι ε, θέμα αποτυχίας έργου. Όχι. Είναι πετυχημένα, απλώς υπάρχουν κάποια οικονομικά σφάλματα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια που έχουν κάνει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γιαλασάντερ που έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και στον κύριο ε, Επίτροπο αλλά και στον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα όσα είπαν. Η αλήθεια είναι η εξή. Εγώ δεν ξέρω. Να κλάψω ή να γελάσω. Γιατί είναι η τελευταία απαλλαγή, όχι μόνο για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και για τον Επίτροπο, τον κύριο Μόιντα. Και αισθάνομαι κάποιο εκνευρισμό, για να μην πω πως αισθάνομαι αμήχανα. Συνήθως με τους επιτρόπους, και ακούγεται λίγο αν, ανόητο, αλλά και με τον κύριο Όιτιγκερ κάναμε μια ένθερμη ανταλλαγή απόψεων, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμφανίζεστε ε, εσείς στην συνέλευση της δικής σας πολιτικής ομάδας, ε, κομματικής ομάδας και τόσο δημόσια να παίρνετε το λόγο. Θα μπορούσατε να έχετε πάει ως ιδιώτης. Και ελπίζω πως στη Λισαβόνα θα έρθετε και στη δική μας πολιτική ομάδα να συγχαρείτε ε, το δικό μας υποψήφιο. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πως ένας κώδικας επικοινωνίας και θα πρέπει οι, επιτρε... επίτροποι να δείχνουν και να είναι ανεξάρτητοι πολιτικά και κομματικά. Αυτό πρέπει να σας το πω γιατί πρέπει να σας πω πως μου φάνηκε πως δεν χρειαζόταν να το κάνετε και δεν ήταν και καλύτερη στιγμή. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ε, πλησιάζουν ευρωεκλογέ. Δεύτερον, για μια φορά ακόμα και έχετε δίκιο. ήρθατε να μα δείτε σαν να είμαστε εμεί οι Ήτρε και να μα παρουσιάσετε τι επιτυχίε. Σα ευχαριστώ πολύ και είναι αλήθεια. Θα πρέπει να συγχαρούμε αλλήλω και στα αποτελέσματα να σα πω πω πραγματικά υπάρχουν περιπτώσει για συγχαρητήρια. Αλλά εγώ σα ρωτώ και δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτό με τα ε, έργα και τα project για το βραβείο Νόμπελ και τα υπόλοιπα μας παρουσιάσατε. Αλλά η δική μου ερώτηση είναι εξή. Αυτό το 4,2% σφάλματο. που υπάρχει ακόμα μετά από τα χρόνια και χρόνια που προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, τι σημαίνει. Σημαίνει πως το ποσοστό είναι υπερβολικά υψηλό. Και έχουμε 100 εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν θεωρηθεί σφάλμα. Και δεν μιλώ για τις περιπτώσεις και τις υποθέσεις που πήγαν στην Όλαφ. Και βέβαια, ναι, αυτό το χρήματα που χάθηκαν ενδεχομένω δεν μα επέτρεψε να πάρουμε κάποια άλλα βραβεία Νόμπελ, γιατί δεν έφτασαν τα κονδύλια σε αυτού που θα έπρεπε να φτάσουν. Ή δεν έφτασαν γιατί είχαμε σφάλματα. Οπότε, εντάξει, μια φορά ακόμα μα προσχέζονται επιτυχίε. Εμά το πρόβλημα μα εδώ δεν είναι τα αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι αν οι δαπάνε έγιναν σωστά. Είπατε, έχουμε μία μείωση, ε, αλλή μόνο πια, αλλά σε σχέση με την περασμένη χρονιά πρέπει να σας πω πως είχαμε μια ελάχιστη αύξηση, ένα δεκαδικό αριθμό. Οπότε είναι χιλιάδες, εκατομμύρια ε, εκατομμυρίων ευρώ που έχετε υπό τη διαχείρισή σας και που χάνονται και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Επίσης, και θα ήθελα να πω στο ελληνικό συνέδριο, πρέπει να σα πω πω χαίρομαι που ήρθατε εδώ και επιπλέον που άλλαξε ο τρόπος που ε, ε, στέλνετε την έκθεσή σας, γιατί τουλάχιστον στην τελευταία ε, απαλλαγή στείλατε και κάποιε υποθέσει στην Όλαφ και τις παρουσιάζετε πρώτες, γιατί στα, σε ανακρίσεις νομίζω <laughs> τα πράγματα, ε, καλά δεν ήτανε. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα. Και αυτά τα βλέπουμε και στη σύνυψη. Δεν μπορώ να πρόκειται να μπω αυτή σε λεπτομέρειε για να εξηγήσω ε, όλους τους λόγους όπως έκανα τι πρώτε χρονιές. γιατί τα πράγματα θα χειροτερεύσουν μεταξύ μα. Αλλά να σα πω πω στις απαντήσει και στι αποκρίσει που είχαμε από το ελεγκτικό συνέδριο πια βλέπουμε πω τα προβλήματα είναι πολλά με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο που δεν λύθηκαν τελικά. Γιατί επειδή αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε για το Horizon 2020, θα λυθούν εκεί. Και μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο φέτος πως ούτε εκεί. Και πως ε, το κόστος προσωπικού, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, που λέτε εσείς ότι θα λυθεί. Εντάξει. Και τι θα γίνει. Θα το αλλάξουν αυτό για θα του δίνουν περισσότερε διακοπέ. Αν έχει κόστο προσωπικού, έχει κόστο προσωπικού. Μην μου λε ότι δεν υπάρχει. Εγώ θα συνεχίσω λοιπόν να ζητώ να ε, πληρώνονται. Και ο υπολογισμός αυτών και το κομμάτι που είναι οι υπερορίες, το μισθολογικό κόστο και όλα αυτά, βλέπω πως το θέμα δεν είναι μόνο δύσκολο, αλλά ακατανόητοι οι κανόνες σε πολλέ περιπτώσεις. Για να μην μιλήσω για τις εξηγήσει που λάβαμε, και μιλάμε για πάνω από 20% των συναλλαγών και των πράξεων και έχουμε μία σειρά από φορεί μη Ευρωπαϊκού. και ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκλέτσερ Πολλέ φορέ έχετε ε, επίμονα ζητήσει τι γίνεται με την Ελβετία και φαίνεται πως το όλο θέμα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό. Φτάνουν οι ευρωεκλογέ και πώς θα πάμε. Να πάμε στην προεκλογική εκστρατεία και να πούμε παίρνουμε βραβεία Νόμπελ επειδή εμεί πληρώνουμε. Αν πληρώναμε περισσότερα γιατί δεν είχαμε απάτες και δεν είχαμε σφάλματα, νομίζω ότι θα είχαμε πιο πολλά βραβεία Νόμπελ στις αποσκευές μας να παρουσιάσουμε. Πείτε μου λοιπόν, σε αυτή την τελική στροφή στην οποία έχουμε φτάσει, τι θα κάνετε εσείς έτσι ώστε τα αποτελέσματα που έχουμε να είναι καλύτερα. Γιατί στο Horizon 2020 τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Το είπε το ελεγκτικό συνέδριο και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε βελτιωθεί. Τώρα για την απλούστευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου δώσατε τουλάχιστον τους πίνακες που ε, ζητώ τόσα χρόνια και επειδή εγώ δεν είμαι πολύ καλή στα μαθηματικά, επιτέλους μου δώσατε πίνακες στους οποίους μπορώ να καταλάβω έμεσα κόστη 25%. Εκεί είναι πολύ εντυπωσιακά τα ποσά. Και σε σχέση με αυτή την απλούστευση, να σας πω ότι δεν ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο. Και θα ήθελα να ρωτήσω και το εξή. Στα 10 έργα, τα πιο ακριβά, που πληρώνουμε από το Horizon 2020, έχετε κάτι νούμερα που λέτε 100%. Δηλαδή, γιατί τους πληρώνουμε το 100% και είναι και στρογγυλεμένα τα ποσά, 88 εκατομμύρια κτλ. Για ποιο λόγο αυτοί λαμβάνουν το 100%. Συνήθως σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουμε ε, ένα όριο συγχρηματοδότησης, ακόμα και στην ΚΑΠ. Και μας είπαν πως αυτό είναι και το πρόβλημα, η λύση για το πρόβλημά μας. Εσείς λοιπόν γιατί τους δίνετε το 100%? Γιατί είναι πολύ δαπανηρά αυτά τα έργα, έτσι κι αλλιώς. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όποτε έχω ζητήσει Πολλές φορές δεν μου απαντάτε. Παρόλο που έχω ζητήσει να εντοπίζουμε ανακράτος, γιατί εντάξει, εμείς ξέραμε περίπου ε, προς τα που γέρνει η μπίλια, αλλά ευτυχώς, ευτυχώς μας δώσει τον κατάλογο ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τις περισσότερες ενισχύσεις. Βλέπω τους υπολογισμούς για τα ευρωπαϊκά προγράμματα επιτέλους στην έρευνα. Και αναρωτιέμαι, σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αριστεία. Γιατί νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζόμαστε να έχουμε και δικαιοσύνη γεωγραφική. Είναι απαραίτητο αυτό για τη συνοχή και για να επιτύχουμε περισσότερη ισορροπία. Οι καλύτεροι θα είναι πάντα καλύτεροι ε, διαφορετικά και οι χειρότεροι θα είμαστε πάντα κάτω-κάτω ε, στις επιδόσεις, στην έρευνα. Εντάξει, οι άλλοι δεν έχουμε αριστεία επειδή μας χτύπησε η κρίση. Και τελικά τι κάναμε μέσω κρίσης, βελτιώσαμε αυτούς που τα πηγαίνανε καλά. Τέτοιο επίτροπο όπω εσεί θα έπρεπε να έχει και στην αριστεία καλύτερε επιδόσει. Γιατί το ξέρετε και από τη χώρα σα πω υπάρχει αριστεία παντού. Και δεν είναι δύσκολο να είναι κανεί άριστο στο Κέμβρι, στην Οξφόρδη, στο Imperial, στο Λονδίνο. Χριστέ μου, με τα χρήματα που παίρνουν κάθε χρόνο. Γιατί αν δίναμε τα ίδια χρήματα και στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, και αυτοί εξίσου καλά θα τα κατάφερναν αν έπαιρναν τα δισεκατομμύρια ε, που παίρνουν αυτά τα κολέγια και αυτοί οι φορείς. Εσείς τι κάνετε, έτσι τουλάχιστον στα πλαίσια του 2020, να μειώσετε σε αυτές τις τραγικές ανισότητες. για να μην χρεθεί η ελπίδα και στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο αυτή η έλλειψη ισορροπίας σε γεωγραφικό επίπεδο που είναι τεράστια να βελτιωθεί. Γιατί αυτή είναι η προσθεμένη αξία της Ευρώπης. ότι η καλή είναι καλή το ξέρουμε. Τι θα κάνουμε έτσι ώστε η καλή να είναι άριστη όπως και σε άλλες χώρες. Και αυτό θα δώσει ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία αν το καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Βεβαίω θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω ότι χαιρόμαστε που υπάρχει ένα πρόγραμμα αριστείας. Το πρόγραμμα έρευνα είναι πρόγραμμα αριστείας και όχι πρόγραμμα συνοχής. Ναι, ναι. Σαφώς. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Το πρόβλημα υπήρχε, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Λοιπόν, ο κύριος Επίτροπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια και είναι η τελευταία μου χρόνια που με κατηγορούν ότι μεροληπτώ στα τέσσερα αυτά χρόνια με έχουν καλέσει παντού σε άλλα κόμματα, σοσιαλδημοκράτες κτλ. Κανείς ποτέ δεν με κατηγόρησε για κάτι τέτοιο. Επιτρέψατε μου λοιπόν να νιώσω κάποια έκπληξη με τα σχολεία σας. Τι ξέρετε, έχω πάει και σε ημερίδες άλλων κομμάτων και ο κάθε επίτροπος πηγαίνει στο συνέδριο του κόμματός του. Δεν τρεπόμαστε γι' αυτό. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τα κόμματα. Α, κυρία Γιάλα Σέντερ, έχω συνεργαστεί με τους πάντες εδώ πέρα, με κάθε βουλευτή. Δεν κάνουμε απολύτως καμία διάκριση και ξέρετε ότι ευχαρίστως να πάω στη Λισαβόνα στο συνέδριο των σοσιαλιστών ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως. Οπότε μου προξένησε σε έκπληξη αυτό το οποίο είπατε. Δεύτερον, ε, μου προξένησε σε έκπληξη επίσης το ότι είπατε ότι έχουμε ένα ποσοστό χρηματοδότησης 100%. Ε, νομίζω ότι αυτό το προβλέπει ο νόμος έχουμε 100% πληρώνουμε το άμεσο κόστος και 25% για το έμεσο κόστος. Οπότε έτσι είναι οι κανόνες του προγράμματος, δεν είναι κάτι το περίεργο. Ή το εξαιρετικό μετά ρωτήσατε για την κατανομή ανακράτος μέλος. Αυτό βεβαίως υπήρχε, το έχουμε απαντήσει στις ε, γραπτές ερωτήσεις θα συνεχίσουμε την απλοποίηση σε όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε. Από το 5,6 πέσαμε στο 4% φέτος. Ε, είναι μια μεγάλη βελτίωση. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε ικανοποιημένοι. Έχουμε κάνει ε, πολλή δουλειά όμως. Και νομίζω ότι έχουμε βελτιώσει τα πράγματα στην απλοποίηση. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν ε, κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, ε, αναλαμβάνω και εγώ το δικό μου το μερίδιο της επιτυχίας βεβαίω αυτής ε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το αρνητικό. Already finished. Τελειώσατε κιόλα. Ε, ναι, ναι, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Ε, είμαι εδώ, εδώ και τέσσερα χρόνια και εξηγώ όλα τα βήματα που έχουμε κάνει. Ξεκινήσαμε με ένα πρόγραμμα που δεν ήταν απλό. Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι το πρόγραμμά μας είναι απλούστερο από τα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο. Ο κόσμος αναγνωρίζει το πόσο καλό είναι το πρόγραμμα αυτό έρευνας και επιστημών σε σύγκριση με άλλα προγράμματα. Και βέβαια, ε, κυρία Γιάλα Σέντερ, ε, μιλάω ακριβώς εδώ πέρα για τις περιπτώσεις της επιτυχίας. Ε, Υπάρχει, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που κακολογούν την Ευρώπη. Ε, ας μην το κάνουμε κι εμείς. Η δουλειά μου λοιπόν ως Επιτροπός είναι να αναφέρω ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις. Και ναι, βεβαίως ε, ξέρουμε πως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε καλύτερα και πρέπει να το κάνουμε. Εντάξει, μπορώ να, είμαι πιο, να δώσω μια πιο πολιτική απάντηση, αλλά ε, δεν βρίσκομαι εδώ πέρα από αυτήν την ιδιότητα. Βρίσκομαι εδώ για να σας πω το εξής είναι σήμερα καλύτερη κατάσταση από ό,τι ανέλαβα καθήκοντα το 2014. Ναι, τότε το ποστό σφάλματος ήταν 5,6, σήμερα είναι 4,2. Έχουμε καλύτερα επιστημονικά αποτελέσματα. Ναι. Οπότε, απορώ λίγο με τα σχολεία σας. Ο κύριος Αλαφράγκα. Ε, gracias, señora ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνεδρίο και τον κύριο Επίτροπο που βρίσκεται εδώ σήμερα. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και από πλευράς μου. Πιστεύω ότι ο Επίτροπος ε, δικαιούται να συμμετέχει σε κάποια διάσκεψη πολιτικού κόμματος. Εξάλλου, επτά Επίτροποι και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο κύριος και ο κύριος Χόγκαν, ο κύριος Χάν, όλοι έχουν συμμετάσχει στις αντίστοιχες διασκέψεις των πολιτικών τους κομμάτων. Η τελευταία έλαβε χώρα στη Μαδρίτη. Οι Επίτροποι έχουν τέτοιο δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά τα συνέδρια. Εγώ τρέφω μεγάλο θαυμασμό για τον Ζακ Ντελόρ, ο οποίος ε, πήγαινε στην Σοσιαλιστική Διεθνή. Φυσικά, η Επιτροπή, ξέρετε, είναι και πολιτική, ενώ ταυτόχρονα έχουν ε, αναλάβει όρκους ε, αμεροληψίας τους οποίους σέβονται. Ε, υπό την ιδιότητά τους ως ε, Επιτροπή δεν πάβουν να προέρχονται από πολιτικές οικογένειες ε, με τις οποίες είχαν κάποια δέσμευση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την πραγματικότητα όταν κάνουμε αξιολογήσεις και να είμαστε και δίκαιοι. Και φυσικά δικαιούται και ο Επιτροπός να μας πει ποιες ήταν οι εμβληματικές επιτυχίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του. Καλό είναι που ε, δόθηκαν μεγάλες χρηματοδοτήσεις ε, για τα σημαντικά οικονομικά προγράμματα. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ε, το πρόγραμμα αυτό για την έρευνα και για την νέα έρευνα για τον καρκίνο και είναι σημαντικό που έχει μειωθεί ο συντελεστής φάλματος παρότι παραμένει λίγο υψηλός. Πρέπει να βελτιστοποιήσουμε το κόστος ε, για το προσωπικό και τα βοηθητικά κόστη, να βελτιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Οπότε αυτό που έχω να ρωτήσω είναι δύο πράγματα ουσιαστικά. Πρώτον, κοίταξε το ερωτηματολόγιο. Υπάρχει ένα κομμάτι που αναφέρεται σε πέντε συγκεκριμένε χώρε. Ε, αναφερθήκατε σε αυτό. Ποιο ποσοστό του προπολογισμού ουσιαστικά πάει σε τρίτε χώρε μπορείτε να μας το αναλύσετε και επίσης θα μπορούσατε να μας πείτε για τις υποθέσεις που θα πάνε στην Όλαφ από ό,τι κατάλαβα ε, είναι πολύ σταθερός ο αριθμός των υποθέσεων που εξετάζει η Όλαφ πολύ μικρός 33, 39 μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα παραπάνω για τη μεθοδολογία που ακολουθείτε μετά πώς γίνεται η διαβίβαση στην Όλαφ, ποια είναι η διαδικασία και τέλο, Ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τη ε, συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας από αυτά τα προγράμματα, ποια είναι η εκτιμήσή σας. Η καινοτομία είναι πολύ σημαντική. Και έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε καλά επίπεδα καινοτομία που πράγματι χρηματοδοτήθηκαν μέσω αυτού του προγράμματος. Νομίζω ότι 128 άδειε ευρεσιτεχνία ε, εγκρίθηκαν πέρυσι. Το 79% αν δεν κάνω λάθος ε, προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μόνο 8%. Ε, συγχρηματοδότηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνία από την Κομισιόν. Μπορείτε να μου ερμηνεύσετε λίγο αυτά τα προγράμματα και αυτά τα νούμερα. Όπως βλέπουμε τα θεσμικά όργανα παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και στη χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα, αλλά νομίζω ότι το 8% είναι πολύ χαμηλό. Και κάτι τελευταίο, κοιτάω το σημείο 23. Το συζητήσαμε με την κυρία Γιαλασέντερ, η χώρα μου. Ε, είναι στην πρώτη θέση εδώ ε, μεταξύ των χωρών ε, που εποφελούνται από την έρευνα στη συνδεσιμότητα. Προφανώς ε, με χαροποιεί αυτό. Αλλά αυτό όμως σημαίνει κιόλα ότι θα πρέπει να καταβάλουμε εντονότερες προσπάθειες ώστε να παρέχεται αριστεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να συμμετέχουν όπως αρμόζει. Όλα στη ζωή μπορούν να βελτιωθούν και εμείς θα πρέπει στην προσπάθειά μας εδώ να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας για το μέλλον. Ευχαριστώ. Κυρία Αγιάλα, θέλετε να παρέμβετε εν συντομία. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η πρώτη η οποία αισθάνθηκε έκπληξη. Όχι που συμμετείχατε, γιατί η συμμετοχή δεν είναι πρόβλημα για μένα. Για μένα το πρόβλημα ήταν η δημόσια δήλωση και επειδή σας παρακολουθώ εγώ στα κοινωνικά δίκτυα, ίσως αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα, μου φάνηκε φοβερό που ε, περηφανευτήκατε στα κοινωνικά σας δίκτυα, πως ήσασταν εκεί με κομματική ε, ταυτότητα. Το ίδιο που έγινε με τον κύριο Έτιγκερ ε, δεν έχω πρόβλημα με το να πάτε. Το πρόβλημά μου είναι αυτή η δημόσια δήλωση που κάνατε. Αυτό μου φάνηκε εμένα ε, παράξενο, γιατί πρέπει να είναι κανείς ανεξάρτητος και να φαίνεται. Αλλιώς κάθε φορά ε, που σε κάποιον πετυχαίνει το λαχείο και το λέω αυτό σε εισαγωγικά, σε κάποιες ε, κυβερνήσεις, ε, θα γίνεται το ίδιο. Αυτό ήθελα να σας πω. Το να πάτε, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σαλαφάνκα. Πηγαίνετε, δεν έχω πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Και ο επίτροπο Έτιγκερ ε, το δέχτηκε και είπε δεν ήταν πραγματικά ε, σωστό που ένας Επίτροπος ε, κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί όταν δεν θα είναι 28 και θα είναι 27... δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν μειώσουμε τον αριθμό θα γίνει βατερλό εδώ μέσα στο Συμβούλιο. Και τουλάχιστον τότε δεν θα έχουμε το πρόβλημα ε, της ανεξαρτησίας ή όχι, γιατί ο καθένας θα εκπροσωπεί ε, παραπάνω από μία κυβερνήσεις. Αυτό. Δεύτερον, όντως βελτιωθήκαμε. Αλλά το 2018 έχει στοιχεία ανησυχητικά. Και επειδή περνάμε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στο Horizon 2020, για το λόγο αυτό, ως μέλος της Επιτροπής, όχι ήτρε αλλά κοντ, να κάνω αυτή τη δήλωση και να πω πως έχουμε πρόβλημα γιατί το ποσοστό σφάλματο και το ελεγκτικό συνέδριο που δεν τα πάγω κύριε Μίδας, το είπε το ελεγκτικό συνέδριο που στο κάτω-κάτω μα δίνει αποτελέσματα ε, τα οποία δεν μπορούμε εμεί να ρυθούμε. Και λέει πω, αυξήθηκε από το 16 στο 17 και από το 17 στο 18 δεν είχαμε σημαντική μείωση, τότε ναι, έχουμε πρόβλημα. Και επειδή παίρναμε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στο Horizon 2020, γι' αυτό ανησυχώ. Πολύ σωστά είπε ο κύριο Σαλφρανκά. Ακόμα 6 υποθέσει έχουμε στείλει στην Όλαφ. Έξι επιπλέον ε, με αυτές τις περασμένου, του περασμένου έτους. Οκτώ προσφυγές παραπάνω από το 16. Αυτά είναι τα στοιχεία του Ελληνικού Συνεδρίου, δεν τα έχω πει εγώ. Και η Γενική σας διεύθυνση λέει πως τα πράγματα δεν ε, βελτιώνονται και είναι δικές σας ελεγκτικές υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο ανησυχία για το 2017. Ε, τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα και δεν έχουμε βελτίωση. Και μα λέει το ελεγκτικό συνέδριο που εκεί όπου τα περισσότερα σφάλματα. Οι κανόνε εξακολουθούν να είναι δυσνόητοι και δύσκολο να εφαρμοστούν. Ε, εκεί φοβάμαι πω η κατάσταση δεν είναι καλή. Και γι' αυτό σα ρωτώ. Ε, το πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών, για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί η απλούστευση του 25% με το καταποκοπή, κλείνοντα τα μάτια για έργα στα οποία το 25% μπορεί να είναι 100 εκατομμύρια, ε, δεν νομίζω πως αυτή η απλούστευση θα πρέπει να ισχύσει έτσι, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος πάντα. Οπότε θέλουμε μια ισορροπία στην κατάσταση αυτή, έτσι ώστε να είναι νόμιμο, αλλά να είμαστε σίγουροι πως αυτή η νομιμότητα δεν δημιουργεί ε, αμφιβολίες και δυσκολίες. Λοιπόν, γεωγραφική κάλυψη. Όχι πάντα οι ίδιοι. Όχι πάντα οι ίδιοι πρώτοι. Η γεωγραφική κάλυψη, θέμενη αξία ευρωπαϊκή. Ναι, γιατί κάποιους δεν τους βοηθήσαμε να φτάσουν στην κορυφή του πίνακα του ranking. Γιατί αν πάντα έχουμε τις ίδιες χώρες στην κορυφή του πίνακα, ξέρουμε γιατί γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στον κώδικα συμπεριφοράς των επιτρόπων λέει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν αξίωμα σε εθνικό κόμμα. Και βεβαίως ε, όσο συμβαίνει κάτι τέτοιο ε, υποθέτουμε ότι τήρηται. Έτσι γιατί θα ήταν ε, κάπως ε, περίεργο να γίνεται διαφορετικά και υπάρχει και ένα ζήτημα με την ιδέα της Ευρώπης και βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι τα γνωρίζουν αυτά και έχουν πάρα πολλές πληροφορίες ε, είναι οι επίτροποι και εγώ γνωρίζω βεβαίως αρκετά πράγματα αλλά δυστυχώς δεν με καλούν τα άλλα κόμματα δεν ξέρω γιατί θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη αλλά σαφές είναι ότι χρειάζεται μια και αναμένουμε μια υπερκομματική προσέγγιση εδώ πέρα στις ε, Βρυξέλλες ε, και θα είναι, ε, θα, θα είναι κάπως ανησυχητικό αν ξαφνικά εμφανιστεί η Πορτογαλία στην πρώτη-δεύτερη θέση των δικαιούχων. Όχι, εντάξει, αν είναι σαφές ότι θα υπάρξουν ερωτήσεις. Θα ήθελα τώρα να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. γιατί ο πίνακα αυτό με του μεγαλύτερου δικαιούχου είναι πολύ ενδιαφέρον και το γνωρίζαμε, αλλά όταν το βλέπει κανείς βλέπουμε εντυπωσιακά νούμερα. Ε, ο κύριος δικαιούχο εδώ πέρα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, λυπούμε λοιπόν, έτσι. Οπότε ποιο είναι το σχέδιο, οι Βρετανοί είναι ε, πολύ μπροστά στις, ε, των 10 πρώτων. Υπάρχει βεβαίως και το θέμα των υπολείπων, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένων των, πολιτι... των πολλών ερευνητικών ιδρυμάτων δεν προξενεί έκπληξη αυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο στα 10 πρώτα έχει 4 πανεπιστήμια. Εάν δει κανεί την συμφωνία απόσυρση, ε, ε, θα συνεχιστεί αυτό. Πώς βλέπετε τον ρόλο των Βρετανικών πανεπιστημίων μετά το Brexit. Για εμάς βεβαίως είναι σημαντικό γιατί η έρευνα πρέπει να είναι επιλογή των ε, καλύτερων. Έτσι δεν κάνουμε συνοχή εδώ πέρα. Για την συνοχή έχουμε τεράστια κονδύλια. Αλλά έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε από το να στρώνουμε δρόμους. Οπότε θα, πρέπει να δούμε πώς θα κρατήσουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια χωρίς να επιβραβεύσουμε και όλα στους Βρετανούς για τον Brexit. Το άλλο θέμα αφορά την Ελβετία. Ε, και Ελβετία εκεί πέρα βρίσκονται στον κατάλογο με ένα εκατομμύριο είναι καθαροί ε, δικαιούχοι. Πώς βλέπετε λοιπόν και τον ρόλο της Ελβετίας στο τρέχον και στο μελλοντικό πλαίσιο έρευνας και θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα για τις ε, ροές των κονδυλίων του ορίζοντα 2020 βλέπουμε ότι αυτή η αργή ροή το βλέπουμε και στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα το 7 έχουμε μία άμεση διαχείριση έχουμε επαγγελματίες επιστήμονες γιατί δεν είναι αλλιώς ε, τα πράγματα είναι τεράστια τα Ναι, μάλλον δεν είναι τεράστια τα, τα ποσά. Και έχει πέσει και το ποσοστό επιτυχία, δηλαδή πρέπει να γράψει κανεί περισσότερε αιτήσει ε, για να καταφέρει να χρηματοδοτηθεί. Έχετε λοιπόν τώρα την ευκαιρία ακριβώ για να απαντήσετε. Άσχορθ, Στεχόφσκι και μετά εσεί, ε, κύριε πίτρο. Ρίτσαρτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Αλλά με όλο το σεβασμό, βρισκόμαστε εδώ σε Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και η δουλειά μα σήμερα είναι να επιβλέψουμε τη διαχείριση και τον ελεγχό των δαπανών στον τομέα τη έρευνα και τη ανάπτυξη. Κοιτώντα τα παραρτήματα εδώ και τα παραδείγματα τα οποία έχουν δοθεί, μου έκανε εντύπωση η λεπτομέρεια της παρουσίασης ε, ε, δεν φανταστικά ότι θα έβλεπαν τα ωράρια των υπαλλήλων. Πιστεύω ότι εδώ το, αυτός ο συντελεστής σφάλματος του 4% κάνει έκπληξη. Τόσο υψηλό, άμα δει κανείς τα times, ήταν δει κανείς τα φύλλα, τα ωράρια των υπαλλήλων, μου έκανε εντύπωση πόσο χαμηλό ήταν το επίπεδο. Επίσης, ε, χάρηκα που άκουσα από τους ελεκτές και από την Επιτροπή ότι αναφέρθηκαν σε απλούστευση. Προφανώς το θέμα της διαχείρισης και του ελέγχου είναι να διασφαλίζεται επαρκής έλεγχος ε, της διαχείρισης του προπολογισμού. Αυτό πρέπει να δισταθμιστεί με το συνολικό διοικητικό κόστος. Και αυτό που είναι ποια είναι η προσθέμενη αξία μιας τόσο αναλυτικής ε, εξέτασης των ε, ωραρίων. Μίλησε ο Επίτροπος ε, για ανασχεδιασμό της ε, χρηματοδοτικής διαδικασίας και μίλησε για καταποκοπή κόστη. Τι εννοεί. Πιστεύω ότι σίγουρα αυτό είναι μια καλή οδός να ακολουθήσουμε για λόγους απλούστευσης. Πρέπει να ξανασκεφτούμε λοιπόν ε, με ποιο τρόπο θα υποστηρίζουμε, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την έρευνα και την ανάπτυξη Κανείς δεν το είπε εδώ. Υπάρχει κάποια δυνατότητα να διασφαλιστεί και κάποιο στοιχείο ανταγωνιστικής ε, προσφοράς των ε, ε, διεκδίξεις μάλλον των έργων. Το να ε, πηγαίνουμε να ερευνάμε τα ωράρια των υπαλλήλων μου φαίνεται λίγο λάθος προσέγγιση ε, τις ωρίες των υπαλλήλων. Ο κύριος Στεχόφσκι παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Μας ενδιαφέρει οτιδήποτε αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων όπως και όταν κοιτάμε αυτό το πίνακα αυτό που μου φαίνεται ενδιαφέρον είναι οι διάφοροι έλεγχοι και μετά τα αποτελέσματα αλλά και οι δαπάνες ε, που συνεπάγονται οι έλεγχοι αυτοί όχι μόνο τα αποτελέσματα διότι συχνά το κόστος των ελέγχων μπορεί να υπερβεί τα χρήματα που έχουμε ανακτήσει. Ε, σε έναν έλεγχο, για παράδειγμα, κάποιων έργων ε, αντιληφθήκαμε ότι πρόκειτο απλά για τις συνθήκες εργασίας, για τις δαπάνες προσωπικού, όπου υπήρχαν κενά σε θέματα χρηματοδότησης και οικονομικές πληροφορίες ε, σε σχέση με τη λογιστική που δεν είχαν δοθεί. Τέτοιου είδους ε, κενά υπήρχαν. Καλό θα ήταν να πούμε κάτι και γι' αυτό και καλό θα ήταν επίσης να δούμε όχι μόνο την περίπτωση της Ελβετίας αλλά και της Νορβηγίας. Με ποιο τρόπο επωφελείται η Νορβηγία από την έρευνα και την ανάπτυξη. Τι γίνεται με τα δικαιώματα δημιουργού, με τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Είχαμε και εμείς κάποιες εμπειρίες ε, όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Πώς ε, έχουν αντιγραφεί αυτά σε άλλες ε, χώρες, πώς εγγράφονται εκεί, τι γίνεται με τα δικαιώματα δημιουργού στην Κίνα για παράδειγμα. ή σε κάποιες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν ε, ε, περιθώρια βελτίωσης ε, διότι όταν επενδύουμε τόσα πολλά χρήματα στην έρευνα θα πρέπει να έχουμε και κάποιες απολαβές τουλάχιστον να μην μας κλέβουν να μην χάνεται αυτή η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τα αποτελέσματα και όχι τα ποσοστά σφαλμάτων κτλ. Δεν είναι αυτά τα πιο σημαντικά. Το σημαντικότερο κατά την απόψή μου είναι να μάθουμε κάτι και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε, στους κλάδους της έρευνας και της ανάπτυξης. Κάτι άλλο που μου φάνηκε ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνα συχνά επικεντρώνεται στο βορρά και στη δύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μήπως θα έπρεπε να μετατοπιστεί κάπω προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από τις διάφορες ερωτήσεις ε, που ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα μια ερώτηση του κυρίου Σαλαφράγκα και του κυρίου Σδεχόφσκη για τις ε, τρίτες χώρες και τη σημασία τους. Θα ήθελα να πω ότι η εμπειρία μας ε, με τις ε, τρίτες χώρες ήταν πάρα πολύ θετική Γιατί η επιστήμη σήμερα είναι παγκοσμιοποιημένη. Η Ελβετία, παραδείγματο χάνει, υπάρχει στο πρόγραμμα πλαίσιο 7. Βλέπουμε 4% τη συνολική χρηματοδότηση ε, στον ορίζοντα έχουν ήδη λάβει 2,6, αλλά σαν 2,3 δι. Οπότε όταν δούμε τους αριθμούς η χώρα αυτή δίνει λεφτά και παίρνει λεφτά και κάτι το οποίο ανακαλύψαμε σε τον χρόνο και το είδαμε στον ορίζοντα 2020 είναι ακριβώ ε, αυτή η ανισορροπία. Κάποιοι δίνουν, κάποιοι παίρνουν περισσότερα και κάποιοι λιγότερα από όσα δίνουν. Στην πρότασή μας λοιπόν αυτή θα δείτε ότι το αλλάξαμε αυτό για να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν βγάζουμε κέρδος, αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους, ε, γιατί θα βρούμε έναν ε, τρόπο έτσι ώστε ό,τι δίνουν ε, να το παίρνουν και έτσι θα υπάρχει μια ισορροπία. Και θα πληρώνουν και ένα τέλος διαχείρισης γιατί υπάρχει κάποιο διαχειριστικό κόστος. Αλλά σας λέω ότι ο μόνος τρόπος ε, για να διαφοροποιηθούμε στην Ευρώπη σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου όπως η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι ακριβώς να είναι ανοιχτή η Ευρώπη και να πούμε ότι κάθε χώρα μπορεί να λάβει μέρος γιατί θέλουμε να μοιραστούμε την γνώση μαζί τους. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτές τις διαφορετικές χώρες υπάρχουν διαφορετικών ειδών χώρες. Μιλάμε για το Ισραήλ, την Νορβηγία, μιλάμε για την πρώτη κατηγορία. Μετά υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Ουκρανία, η Τινησία που είναι περισσότερο θέμα επιστημονικής διπλωματίας. Αλλά περίεργως και εκεί πέρα υπάρχουν εκπληκτικά πράγματα. Ήμουν στην ε, Αρμενία όπου βλέπουμε πραγματικά ε, ένα εκπληκτικό πρόγραμμα μετά το σχολείο στο οποίο εκπαιδεύονται τα παιδιά στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και είναι τόσο καλό το σχολείο ώστε αποφασίστηκε να μεταφερθεί το έργο αυτό και στο Παρίσι. Οπότε μαθαίνουμε πολλά από τις τρίτες χώρες. Και μετά υπάρχει αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Σαλαφράνκα για το θέμα της απάτης ε, το οποίο πραγματικά με κάνει να μην κοιμάμαι. Στηρίζουμε πλήρως ε, το έργο του Όλαφ είχαμε ακριβώς την αύξηση αυτών των περιπτώσεων και μπορώ να σας πω ότι καθόλου δεν ε, ε, επαναπαυόμαστε, μπορεί να στα πει και ο Γενικός ε, Διευθυντής. Αυτές τις ημέρες επεξεργαζόμαστε ακριβώς την στρατηγική καταπολέμηση της απάτης και πραγματικά το πολεμάμε όσο μπορούμε, αλλά πάντα θα υπάρχει απάτη, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Ε, βεβαίως πρέπει να έχουμε το σύστημα, τα νέα πληροφορικά εργαλεία. Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε ως μια συστηματική αύξηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θέλω να πω. Μετά για την ε, καινοτομία. Γεγονός είναι ότι η πλευρά του δημοσίου δεν τα πήγαινε τόσο καλά όσο η πλευρά του ιδιωτικού τομέα στο θέμα των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πώς μπορούμε λοιπόν ακριβώς ε, να τους βοηθήσουμε και τους ε, δύο, γιατί ακριβώς δεν είναι το θέμα να έχουμε μόνο τον δημόσιο τομέα, αλλά να συνεργάζονται. Μετά. Η κυρία Γιάλα Σέντερ μας μίλησε για το επίπεδο του ποσοστού σφαλματος. Κοιτάξτε, εγώ είμαι μηχανικός. Όλη μου τη ζωή ασχολούμαι με αυτά τα νούμερα και θα ήθελα ο κ. Μπένικ Μαέρ να μας πει ποια είναι η διαφορά μεταξύ 4,1 και 4,2. Δηλαδή, ήμασταν στο 5,6. Πέσαμε στο 4,1. Και μετά φέτος από 4,1 στο 4,2. Δηλαδή οποιοδήποτε μαθηματικός θα σας πει ότι δεν υπάρχει διαφορά ε, στο 4,1 με 4,2. Η τάση είναι πτωτική. 4,1 ε, με 4,2 είναι απελταία η διαφορά. Και μετά είπατε και κάτι άλλο, κυρία Γιάλα Σέντερ, για τις χώρες που πρέπει να βοηθήσουμε. Το έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ. Έχουμε το πρόγραμμα του ορίζοντα στην Ευρώπη για το πώς θα διαδοθεί η αριστεία. Λοιπόν, όταν ήρθε η πρόταση στο Κοινοβούλιο, θυμάμαι ότι το είχαμε συζητήσει. Πήγαμε από ένα ποσό το οποίο δεν ήταν καν ένα δισεκατομμύριο στα δύο δισεκατομμύρια για τη διεύρυνση. Το άλλο το οποίο είδα αυτά τα τέσσερα χρόνια είναι ότι πολλά από αυτά τα μεγάλα ιδρύματα, αν πάμε σε ένα ίδρυμα το οποίο είναι πάρα πολύ καλό στην Γερμανία ή στην Βαρκελόνη που δώσατε το παράδειγμα ή στο Ενωμένο Βασίλειο, πολλοί από τους επιστήμονες αυτούς δεν είναι από αυτή την περιφέρεια ή τη χώρα, στο Imperial, στο Λονδίνο. 1500 άνθρωποι, ε, προσωπικό, καθηγητές δηλαδή, δεν είναι Βρετανοί πολίτες. Είναι από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Απλά θεωρούν ότι είναι τόσο καλό αυτό το ε, πολυτεχνείο, όπως θέλουν να πάνε εκεί. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη και πρέπει ακριβώς ε, να βοηθήσουμε αυτά τα ιδρύματα να γίνουν καλύτερα. Γιατί λοιπόν ε, κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες για τη έμβριση. Αν καταφέρουμε το Max Planck να πάει στην Πορτογαλία όπως έκανε το Ινστιτούτο Fraunhofer στο Πανεπιστήμιο του Οπόρτο που άνοιξε εκεί πέρα ε, μια θηγατρική. Τότε συνεργάζονται τα δύο ιδρύματα και έχουμε ανθρώπους Γερμανούς που πάνε στο Πόρτο και ανθρώπους από το Πόρτο που πάνε στη Γερμανία. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε πιο πολύ ακριβώς σε αυτή την διεύρυνση και στην διάδοση της αριστείας. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να σας πω. Εμείς πάντα λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και ακριβώς υπάρχει αυτό το οποίο δημιουργήσαμε η σφραγίδα της αριστείας έτσι ώστε κάποιος ο οποίος έρχεται στον ορίζοντα 2020 αλλά δεν έχει την, δεν παίρνει τη χρηματοδότηση να την πάρει τελικά από τα ε, διαρθρωτικά ταμεία. Ε, δεν είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά αλλά τώρα γίνεται καλύτερο. Και τώρα διαδίδεται ακριβώς αυτή η σφραγίδα της αριστείας στο πρόγραμμα Marie Curie και σε άλλα. Αυτό ήθελα λοιπόν να αναφέρω. Μετά, κυρία Γκρέσλε, μας ρωτήσατε για τους κορυφαίους δικαιούχους και το Ηνωμένο Βασίλειο, το Brexit και τον ρόλο του Brexit. Ξέρετε, όπως ξέρετε εγώ θεωρώ ότι όποια λύση βρούμε το ερευνητικό πρόγραμμα χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται το ερευνητικό πρόγραμμα. Θα βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που θα περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς εδώ σε αυτή την αίθουσα. Υπάρχει το θέμα της γενικότερης συμφωνίας, αλλά αν δει κανείς ε, τους αριθμούς βλέπουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι θεμελιώδης εταίρος και όταν μιλάω με τους ερευνητέ του Ηνωμένου Βασίλειου ξέρουν πως και εμείς είμαστε θεμελιώδης εταίρος. Δεν θα είχαν το επίπεδο επιστημονικής έρευνας που έχουν χωρίς εμάς και αντιστρόφως. Οπότε εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και είμαστε σαφείς ακριβώς για αυτές τις συνδεδεμένες χώρες. Δηλαδή πριν είχαμε Διαφορετικού τρόπου ε, για να συμμετέχουν. Τώρα είναι πιο απλό. Αν θέλει κάποιο να είναι συνδεδεμένο, έρχεται, πληρώνει το κομμάτι που του αναλογεί, πληρώνουμε ε, το κομμάτι που μας αναλογεί και ε, πληρώνουν και το κομμάτι της διαχείρισης, κάποια τέλη. Επίσης, αν θέλετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα βασίζεται στην αριστεία, κατά οποίο θέλουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες οι οποίες δεν μπορούν να, ανέβουν, αλλά να παραμείνει και ο τομέας της αριστείας. Αυτό κάνει τη διαφορά. Έτσι ακριβώς ε, κερδίζουμε τα Νόμπελ και τα έργα εκείνα τα οποία πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι έτσι θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε ένα υψηλότερο σωστό επιτυχίας γιατί ακριβώς ήταν τόσο επιτυχημένο το πρόγραμμα ώστε δεν είχαμε λεφτά για όλα τα καλά έργα που είχαν προταθεί. Το δεύτερο είναι πώς μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο με τα διαφορετικά ταμεία γιατί εάν δεν βρούμε τις ε, διόδους από εκεί, ε, δεν θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή αν έχουμε ένα έργο κάπου σε κάποια περιφέρεια της Ισπανίας, ε, έρχεται σε εμά και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το στηρίξουμε, θεωρώ ότι θα πρέπει να το στηρίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία και να συνεργαστούμε για κάτι τέτοιο και αυτό θα μας ε, επιτρέψει να έχουμε και ένα υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Πράγμα το ποσοστό επιτυχίας είναι πρόβλημα εδώ, το παραδέχομαι. Δηλαδή ο κόσμος λέει γιατί να πάω αν είναι τόσο χαμηλό. Αν έχουμε λοιπόν 100 δισεκατομμύρια θεωρώ ότι θα έχουμε ένα υψηλότερο ποσοστό ε, επιτυχίας. Ξέρετε έχουμε την πρώτη και τη δεύτερη φάση, δύο φάσεις για να φτάσουμε στην επιχορήγηση και Βεβαίω αυτό αποφάρινε τον κόσμο γιατί πήγαινε στην πρώτη φάση, ε, ήταν κάτι το συναρπαστικό και μετά δεν έπαιρναν την επιχορήγηση στη δεύτερη φάση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και μετά, ε, κύριο Άσχουρθ, τον ευχαριστώ για τα σχόλιά του. Πραγματικά τα σχόλιά σας ε, μας επαναφέρουν στην ουσία της συζήτησης. Θέλουμε λογοδοσία και κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό αλλά εδώ μιλάμε για λάθη λάθη ας τα πω ειλικρινή λάθη τα περισσότερα από αυτά είναι ειλικρινή λάθη ε, κάποιοι δεν υποβάλλουν το σωστό έντυπο για τα έξοδα ταξιδίου κάποιος προσπαθεί να υπολογίσει τις ώρες με λάθος μέθοδο και ε, αν δείτε το πού είναι αυτά τα σφάλματα. Πολλά από αυτά είναι οι νέοι συμμετέχοντες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε μια ιδέα θα μπορούσε να είναι για να έχουμε 0% σφάλμα να πούμε κοιτάξτε όσοι δεν έχουν λάβει μέρος στο παρελθόν να μην ε, ξαναέρθουν. Αυτή είναι και αυτή μια λύση, αλλά δεν το θέλω αυτό. Θέλουμε καινούριου ανθρώπου ε, που δεν είχαν λάβει μέρο στο παρελθόν, αλλά όπως είπε και ο κύριο Άσουαρθ, ε, έρχονται, κάνουν λάθη ε, στη γραφειοκρατία. Αλλά καμιά φορά έχουν εντύπωση ότι τα κοιτάμε και λέμε όλοι αυτοί προσπαθούν να μας εξαπατήσουν. Όχι. Υπάρχει ένα έργο εδώ το οποίο ήθελα να αναφέρω. Το έργο αυτό στην ε, Τανζανία. Υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα με το κόστος ε, και τα λογιστικά δεν τα έκανε σωστά. Αλλά αυτό το οποίο έκανε ο κόσμο στη γενική διάθεση ήταν να πάει στου ανθρώπου αυτού, να του ακολουθήσει. Πήγαιναν από χωρίου ει χωρίων, βοηθούσαν τον κόσμο και βοηθούσαν τον κόσμο. Λοιπόν, εάν ρωτήσετε του συναδέλφου που ήταν στην Τανζανία και του είδανε, ε, λέγανε Μα κάνανε φοβερή δουλειά. Αλλά μετά ε, έκανα λάθος στα λογιστικά. Αυτό ε, δεν μπορεί να... εντάξει. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να βλέπουμε σφαιρικά την εικόνα. Δηλαδή, Μια φορά ο κόσμο που κάνει λογιστικά λάθη, αλλά κάνει πολύ καλά και αξιόλογα έργα που αλλάζουν τι ζωέ ε, των ανθρώπων. Ήθελα λοιπόν να το αναφέρω αυτό. Και η κυρία Σουόρθ, αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι ακριβώ να έχουμε κάποια ποσά κατά αποκοπήν. Και άρα θεωρώ ότι Θα σας ε, στείλω την απάντηση για το πόσο λαμβάνει κάθε χώρα, συνδεδεμένη και τρίτη χώρα. Δεν τα έχω τώρα πρόχειρα, δηλαδή ξέρω για την... Έχω εδώ την Ελβετία, το Ισραήλ, Νορβηγία δεν το έχω πρόχειρο, θα σας τα στείλω σε εσά και τον κύριο Σαλαφράγκα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, πάρα πολύ ε, και για τις ερωτήσεις για τη συμμετοχή στα κομματικά συνέδρια. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό σήμερα να υπάρχει και αυτή η κοινωνική συμμετοχή. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να δαιμονοποιούμε πολιτικά κόμματα. Αυτό θα είναι κακό και για τη δημοκρατία. Πρέπει να σας πω, ναι, ναι, ευχαριστώ δεν έχω πρόβλημα με, την συνάντηση, με τις συναντήσεις των επιτρόπων που είναι δημόσιες. Το πρόβλημά μου είναι οι κρυφές, τις οποίες δεν ξέρουμε. Έτσι. Χωρίς να, να αφορά εσάς, αλλά είναι σαφές ότι γίνονται σχέδια για το μέλλον και πιθανώς και συμφωνίες. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, αλλά αυτό το οποίο δεν βλέπουμε. Σας ευχαριστώ για την συζήτηση και για τις επιτυχίες. Έχω μία ερώτηση. Υπάρχει τώρα μία συζήτηση και στην Γερμανία για την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως εκεί πέρα παίζουν ηγετικό ρόλο οι Αμερικανοί, το Google, ε, το ένα τρίτο των ε, αποφύτων κατευθύνονται προς τα εκεί και ίσως και περισσότερο. Και βεβαίως το θέμα είναι η υπολογιστική δυνατότητα και ίσως η Ευρώπη εκεί πέρα να μην είναι τόσο ε, μπροστά. Οπότε μπορείτε να μας πείτε εκεί πέρα τι χρήματα απαιτούνται για να δημιουργηθούν αυτές οι υπολογιστικέ δυνατότητες και να συζητήσουμε το εξής ζήτημα. Έρχονται τώρα καθηγητές που λένε πρέπει να μας χρηματοδοτήσετε και τα λοιπά, αλλά μετά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εμεί ιδιωτικά τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά και την δική σας για την ιδιωτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών ποια είναι εκεί η άποψή σας ε, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Είναι σημαντικό νομίζω να μας ενημερώσετε γι' αυτό. Εκτός μικροφώνου. Uh, uh, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως δύο σημεία πρέπει να υπογραμμίσουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά για το επιστημονικό μας μέλλον. Καταρχήν η τεχνητή νοημοσύνη και δεύτερον η κβαντική τεχνολογία. Για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσαμε να δείξουμε εμείς το δρόμο. Πρώτον, κανονιστικό πλαίσιο. Σήμερα συμφωνούν όλοι πως αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο στην κανονιστική διαδικασία θα ηγηθούν της όλης τεχνητής νοημοσύνης. Σε κάποια κομμάτια του πλανήτη θεωρούν την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα εργαλείο κρατικής ε, παρακολούθησης. Αυτή δεν είναι η δική μας άποψη. Εμείς μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το κανονιστικό πλαίσιο που θα διαμορφώσει τεχνητή νοημοσύνη υπέρ της ανθρωπότητας. Και αυτό θα πρέπει να είναι το δικό μας όρομα. Θα πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να μας στηρίζει, να μας συμπληρώνει ως ανθρώπινα όντα. Το πρώτο λοιπόν είναι ποιες είναι οι πολιτικές αποφάσεις που έχουμε λάβει στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου, γιατί αυτό είναι για το μέλλον, έτσι ώστε να κάνουμε περισσότερα. Για να μπορούμε η τεχνητή νοημοσύνη να μας υπηρετεί στο μέλλον. Αν τα καταφέρουμε, τότε οι επιστήμονες στην Ευρώπη θα ακολουθήσουν αυτή την τάση, γιατί οι επιστήμονες περιμένουν ακριβώς για αυτή την πολιτική απόφαση. Το δεύτερο είναι τα δεδομένα. Τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια τεχνολογία γενικής κατεύθυνσης, όπως και η δημοκρατία είναι μια τεχνολογία γενική. Τα δεδομένα λοιπόν Ξέρετε, μέσα σε τέσσερα χρόνια που είμαι επίτροπος, η πρώτη φορά που άκουσα τόσα πολλά θετικά για την Ευρώπη στην ε, αμερικανική τηλεόραση, ε, στο Fox News και στο CNN, ήταν η προστασία των δεδομένων. Όταν ο Tim Cook και ο Bill Gates έρχονται και λένε «Αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε». Γιατί τα δεδομένα είναι κομμάτι της αξιοπρέπειάς μας. Και αν θέλει κανείς να αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι μια γενική τεχνολογία η οποία βασίζεται σε δεδομένα τα οποία δεν είναι προκατελημένα. Είναι ε, δεδομένα τα οποία έχουν αποθηκευτεί με προσοχή. Αν μου πείτε λοιπόν αυτή τη στιγμή ποιος ηγείται στο κανονιστικό πλαίσιο για να δώσουμε το μέλλον, τότε ναι, είναι η Ευρώπη και αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό το οποίο δεν κάνουμε είναι το επενδυτικό κομμάτι και το είπατε προηγουμένως. Γιατί όταν έχει κανείς εταιρείε όπως η Apple ή η Google, οι οποίες όπως εχουν έχουν αξία 1-3 για παράδειγμα, μπορούν να επενδύσουν περισσότερα από ότι οι κυβερνήσεις. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να συνεχίσουμε να επενδύουμε, γνωρίζοντας όμως ποια είναι τα ωριά μας. Ο Tim Cook, όταν έρχεται εδώ γνωρίζει πως Ό,τι και να κάνουμε, εμείς θέτουμε τα πρότυπα στην Ευρώπη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο και για το μέλλον, όπου, το, όπου οι ευρωβουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την όψη του μέλλοντος. Όλοι έχουν στραφεί προς την Ευρώπη και είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί υπάρχει η ευρωπαϊκή επιρροή στο θέμα αυτό. Αυτή τη μάχη δίνουμε. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε κάποιες ε, κατευθύνσεις μέσα στο Horizon 2020 που θα μας οδηγήσουν εκεί. Σκέφτομαι και τις κβαντικές τεχνολογίες. Γιατί έχουμε από τη μία την νοητή τεχνητή νοημοσύνη, με συγχωρείτε, και αφετέρου την κβαντική τεχνολογία που είναι πολύ πιο σημαντική γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα πει ότι έχουν οι αλγόριθμοι στα δεδομένα. Η κβαντική τεχνολογία αλλάζει τελείως το μοντέλο που ακολουθούμε. Είχατε τη φυσική για τα μεγάλα αντικείμενα. Τραπέζι, ποτήρι, ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν, σύμφωνα με την κλασική φυσική. Όταν μιλάμε όμως για πάρα πολύ αντικείμενα, ο τρόπος που συμπεριφέρουν είναι τελείως διαφορετικός από αυτά τα οποία φαίνονται. Αυτή είναι η κβαντική τεχνολογία και φυσική. Και λυπάμαι που θα αναφερθώ πάλι σε μία από τις επιτυχίες μας, αλλά στο Delft που δεν είναι μακριά από εδώ, έχουν έναν από τους πρώτους κουβαντικούς υπολογιστές και το άτομο εκεί μου έλεγε «Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που δεν μπορείτε να τα λύσετε σήμερα. Μπορεί να έχει κανείς τον πιο γρήγορο υπολογιστή και με την ε, υψηλότερη απόδοση. Αλλά κάποια προβλήματα δεν λύνονται μέσω ταχύτητας. Λύνονται με διαφορετικό τρόπο που δεν έχει να κάνει με πολύ γρήγορους υπολογισμούς γιατί έχει σωματίδια τα οποία μπορεί να είναι δύο σωματίδια μαζί αυτό είναι ο ορισμός του ε, κβαντικού είναι τα ε, ελάχιστο μεγέθους ε, σωματίδια που έχουν διαφορετικές συμπεριφορές παράλληλα δηλαδή μπορεί να είναι 0 ε, και 1 οι τιμές τους μπορεί να είναι ζωντανά ή ε, μη ζωντανά. Είναι πολύ δύσκολο για τη δική μας ανθρώπινη ευθεία να το καταλάβουν αυτό. Όταν όμω είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία σήμερα είναι δυσεπίλητα ή άλυτα, γιατί κάποιες εξισώσεις σήμερα χρειάζονται όχι μόνο να λυθούν με ταχύ τρόπο, αλλά με σωματίδια τα οποία συμπεριφέρονται με ε, ανακόλουθους τρόπους. Αν έχουμε λοιπόν το συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και κβαντική τεχνολογία θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και η νέα γενιά θα λέει πώς ήταν η ζωή πριν το ίντερνετ και σε 50 χρόνια θα λένε πώς είχαν υπολογιστέ που δεν ήταν κβαντική τεχνολογία, Πολύ σημαντικό σημείο αυτό για μας. Μάλλον δεν θα έχουμε τα ίδια χρήματα που έχουν οι μεγάλες εταιρείες στη διάθεσή μας, οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι, αλλά έχουμε τους επιστήμονες και γι' αυτό πρέπει να συνεχίζουμε να τους φροντίζουμε επενδύοντας σε αυτούς και στα προγράμματα επιστήμης. Thank you very much. Um, το ελεγκτικό συνέδριο παρακαλώ. Όσον αφορά την ερώτησή σας, ε, τι θα κάνουμε με το ιδιωτικό και το δημόσιο κέρδος από κάποια έργα Πρέπει να σημειώσουμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το EIT, το οποίο ε, ενισχύει την καινοτομία στη Βουδαπέστη, φέρνει έργα στην αγορά και αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Το MIT είναι εντελώς ιδιωτικό ενώ στην Ευρώπη το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινοτομίας και Τεχνολογίας είναι ε, ε, δημόσιο και αυτό κάνει διαφορά. Δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Η μία είναι ότι οι ικανότητες ε, των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλίων για να μπουν και να το στην αγορά είναι αδύναμες. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινοτομίας και Τεχνολογίας, το EIT, προσπαθεί να επιφέρει κάποια βελτίωση. Το ελεγκτικό συνέδριο τώρα ξεκινά έναν έλεγχο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία. Σκοπό είναι να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για το πώ λειτουργούν τα πράγματα στην Ευρώπη, τι βοηθά την Ευρώπη. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι επιτυχής startup στο στάδιο που αναφέρατε όταν υπάρχουν τέτοιες, ε, τι γίνεται, οι μεγάλοι τις εξαγοράζουν για εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή όπου παγκοσμίως η ανάπτυξη της καινοτομία είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά και με κάποια χαρακτηριστικά κάπως ε, επικίνδυνα για την Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι έχουμε το ενημερωτικό μας δελτίο και την ειδική μας έκθεση για την απλούστευση. Σε αυτές τις εκθέσεις έχουμε συμπεριλάβει ε, πολλές πληροφορίες, έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στις περιφερειακές διαφορές οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες, ε, μας ανησυχούν. Από τη μία πλευρά υπάρχει ισχυρή βούληση διάδοσης ε, ε, της γνώσης και της έρευνας και της ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτές οι διαφορές όσον αφορά τη διάδοση ε, δεν έχουν επιτευχθεί. Το ορίζοντας 2020 αφορά την αριστεία όπως είπατε. Υποτίθεται ότι είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει να διαδοθούν περισσότερο τα ευρωπαϊκά έργα Στο ενημερωτικό μας έγγραφο και στην ειδική μας έκθεση λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ του ορίζοντα 2020 και των διαρθρωτικών ταμείων. Υπό ποια έννοια ότι για να υποστηριχθεί η ιδέα της αριστείας θα πρέπει να καλυφθεί το κενό μεταξύ, η διαφορά μεταξύ των χωρών που είναι πιο ανεπτυγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες στον τομέα αυτών. Και με την προσέγγιση του ορίζοντα 2020 πιστεύω ότι θα μπορέσουν να επιφοληθούν και άλλες χώρες. Στις χώρες με πιο αδύναμες επιδόσεις ε, εντός του ορίζοντα 2020 το πρώτο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι το χαμηλό ποσοστό αιτήσεων. Όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε, ένας από τους κινδύνους των προγραμμάτων αυτών είναι το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας. Θα έλεγε κανείς ότι το ίδιο το πρόγραμμα ορίζοντας 2020 έχει χαμηλή επιτυχία. Ελάχιστοι έχουν ετηθεί ε, κονδύλια από τον ορίζοντα 2020. Από την άλλη όμως το κόστος ε, για επιμέρους ε, ερευνητές ε, όταν ετούνται για κονδύλια είναι εξαιρετικά υψηλό. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι σε πολλές χώρες το ποσοστό αιτήσεων, ο αριθμός των αιτήσεων είναι πολύ χαμηλός. Δεύτερον, το ποσοστό επιτυχίας επίσης είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό μεταφράζεται και σε χαμηλό ποσοστό συμμετοχή σε ορισμένε χώρε. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σε κάποιο βαθμό προγράμματα όπω το πρόγραμμα Πλαίσιο 7, το Ορίζοντα 2020 και το Horizon Europe που θα έρθει στο μέλλον, ε, κάνουν κάποιε προσπάθειες ε, το καθένα με τον τρόπο του, για να γίνει κάπως αποτελεσματική η έρευνα. Ο Επίτροπο Βέντα ε, με προκάλεσε κάπως να αναφέρω τη σπουδαιότητα μεταξύ των συντελεστών σφαλμάτων 4,1 και 4,2 πέρυσι για το 2016 και το 2017 και σε σχέση με το φετινό έτος. Σύμφωνα με τη δική μας μεθοδολογία συμπεραίνουμε ότι όπως είπα στην εισαγωγή μου παρατηρείται καθοδική τάση ε, του συνολικού συντελεστή του κεφαλαίου 5 του συνολικού συντελεστή σφάλματος. Το 2014 ήταν 5,6 και τώρα είναι λίγο παραπάνω από το 4, οπότε ε, μειώνεται. Αυτή η τάση αντικατοπτρίστηκε από την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και τις παρατηρήσεις που αφορούν προγράμματα όπως τον ορίζοντα 2020. Στατιστικά όμως θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι η διαφορά μεταξύ του 4.1 και του 4.2 δεν είναι σημαντική. Σημαντική αλλαγή θα ήταν μια αλλαγή τουλάχιστον του 1%. Uh, the change from uh, Μεγάλη ε, αλλαγή μεταξύ του FP7 και του Horizon 2020 δυστυχώς είναι ότι ο συντελεστής σφάλματος μας δείχνει ότι οφείλεται στο το, το 2 τρίτα των συναλλαγών είναι από το προηγούμενο ε, ε, πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο και τέλος η εισηγήτρια. Παρακαλώ, εν συντομία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήταν μια ανταλλαγή απόψεων πολύ ενδιαφέρουσα γιατί μάθαμε πολλά και καινούργια τα οποία είναι χρήσιμα για την εκθέσή μας. Λυπάμαι. Λυπάμαι που όταν έκανα την πρώτη μου παρέμβαση γιατί αναφέρθηκα σε αυτά που με ανησυχούν και δεν μ' αρέσουν, ζήτησα αυτή αντιστοιχεί στο Horizon 2020. Για να έχουμε κι εμείς ε, ε, κάποια γνώμη και ένα τρόπο να λύσουμε ε, τα προβλήματα τα οποία δεν μπορέσαμε να λύσουμε μέχρι σήμερα στο Horizon 2020. Και επιτέλους, στη δεύτερη απάντηση, μας έδωσε το κλειδί για κάποιες από τις λύσεις που θεωρώ ότι είναι θεμελιώδεις. Και έχετε δίκιο, το προσωπικό αυτών των φορέων που είναι πολύ συχνά άνθρωποι από την Ευρώπη, αλλά και από τρίτες χώρες. Αλλά γιατί πάνε εκεί. Είναι ακριβώς το γεγονός ότι βρίσκεται στους καταλόγους αυτών των ε, άριστον επιδόσεων, γιατί έχουν χρηματοδοτηθεί τόσο πολύ. Ε, νομίζω το Cambridge και η Οξφόρδη μετά την, ε, το Brexit θα γίνουν τρίτη χώρα και θα δούμε τι θα γίνει τότε και αν θα χρηματοδοτούνται έτσι. Τώρα, θα πρέπει η προστιθέμενη εξή αυτή να πάει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε θεσμούς αριστείας που θα είναι στο, στην κορυφή των καταλόγων των άριστων και αυτό θα φέρει τη διαφορά. Και έχουμε ερευνητέ που θα πηγαίνουν από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αλλού και με αυτό συμφωνώ απόλυτα αλλά να πηγαίνουν σε αυτούς τους φορείς που δεν θα πρέπει να είναι Max Planck το όνομά του, αλλά θα μπορεί το όνομα να είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα και εσείς έχετε κάποιον ε, Πορτογάλο ποιητή όπως ο Καμόες ή μεγάλο ερευνητή για να δώσουμε ένα όνομα το οποίο θα είναι πορτογαλικό και όχι γερμανικό πια. Και εγώ θα ήθελα να έχω ένα άριστο πανεπιστήμιο, όχι μόνο αυτό της Βαρκελόνης στο πανεπιστήμιο, αλλά στη ε, Σαραγώσα, στη Βιτόρια, στη Μαδρίτη, που να είναι περίφημο γιατί όσο τα έχουμε στην επικράτειά μας θα ποτίσουν και τους υπόλοιπους. Γιατί όπως με, τα, με τους ε, Ολυμπιακούς Αγώνες, αν δεν έχει κανείς τη βάση δεν μπορεί να ε, τους οργανώσει. Και νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη ε, να κάνει ό,τι μπορεί. Ευχαριστούμε. Φτάσαμε στο τέλος της ακρόασης. Ευχαριστούμε και Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία, αλλά πιστεύω ότι θα ξαναειδωθούμε, αν δεν κάνω λάθο. Ε. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε λοιπόν στο σημείο 15 της ημερησίας διάταξης, γνωμοδότηση για την έκθεση της ΑΦΚΟ για τον άσκηση πολιτικού ελέγχου επί της Επιτροπής. Ο κύριος Στεχόφσκι είναι ο εισηγητής. Ε, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ε, ευχηθώ να ξαναγυρίσετε. Ε, μία ώρα μας μένει και να σας πω πως θα μιλάμε μόνο τσεχικά σε αυτή την αίθουσα. Εντάξει, βόμβο η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας είναι της ΑΦΚΟ και είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν, εάν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση η οποία θα είναι σοβαρή για τις μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα συνεχίσω, θα, σας αφήσω να αποχαιρετήσετε τον Επίτροπο και μετά ξαναπούμε στη συζήτηση. Ωραία λοιπόν, τώρα που καθίσατε, αν μιλάμε για σοβαρή μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει καταρχήν να κάνουμε το εξής. Να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα που μπορούμε να πετύχουμε. Check effect πρέπει να δούμε πώς μπορούμε εμείς να ελέγχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί επικρίνουμε πολύ συχνά τα κακό κείμενα, αλλά ορισμένες φορές υπάρχει και ένα πρόβλημα ε, στο γεγονός. Κανείς δεν προσπαθεί να αλλάξει, να αντιστρέψει, να καλύψει τα κοινά. Κανείς δεν προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε και ο, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ακριβώς να ασκεί αυτό το δημοκρατικό έλεγχο ε, στα υπόλοιπα ε, όργανα. Ε, είναι σημαντικό για την ίδια τη δημοκρατική διαδικασία και η ευθύνη αυτή βαρύνει εμάς, την έχουμε αναλάβει λόγω των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι μας εξέλεξαν. Και υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε κάποια κράτη-μέλη, όπου ο ρόλος ο, ελεγκτικός του Κοινοβουλίου είναι λίγο αποτελεσματικός και όχι αρκετά αναπτυγμένος. Αυτό βέβαια συνήθως ε, φαίνεται όταν απλώς υπερψηφίζουν νομοσχέδια, ε, ε, γνωμοδοτούν απλώς χωρίς να μπορούν να ελέγξουν τις κυβερνήσεις. Εμείς είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε, έχουμε τις αρμοδιότητες που μας έχουν ανατεθεί είναι σημαντικό και πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί ο προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και να δούμε οι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί. Ελέγχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ένα ισχυρό εργαλείο το Ελεκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ένα ρόλο το οποίο καλούνται να εκτελέσουν. Και αν χρειαστεί, μπορούμε να χτυπήσουμε και το χέρι στο τραπέζι. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα όργανα τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις μας. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το Συμβούλιο, για παράδειγμα, για διάφορα χρόνια δεν έχει λάβει απαλλαγή. Μήπως πρέπει να τους πιέσουμε παραπάνω γιατί η διαδικασία απαλλαγή είναι ένα κατασταλτικό δημοκρατικό έλεγχο που αποτελεί κομβικό σημείο του δημοσιονομικού συστήματο που έχουμε με συγκεκριμένε συστάσει στα πλαίσια του ευρωπαϊκού θεματολογίου. Θα επιμείνω σε αυτό. Καταρχήν είναι απαραίτητο να φανούμε πολύ προσεκτικοί τη στιγμή που δίνουμε την απαλλαγή. Έτσι ώστε οι πολίτες μας να κατανοούν πως το Κοινοβούλιο έχει ακριβώς και ασκεί αυτή την αρμοδιότητα ελέγχου. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κάποιων εκπροσώπων των κρατών μελών θα πρέπει, και το έχουμε πει πολλές φορές, να παρεμβαίνουν και να μην κάνουμε το ίδιο που είπε η κυρία Κρέτσου και να λέμε πως ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όχι. Στην Τσεχία έχουμε μια ωραία παροιμία την οποία δεν θα σας πω, γιατί δεν θα καταφέρουν να την μεταφράσουν οι διερμηνείς, αλλά να σας πω πως η απαλλαγή θα πρέπει να μπορεί να συνοδεύεται και από κυρώσεις σε περίπτωση που για παράδειγμα δεν σας έχει ε, ε χορηγηθεί απαλλαγή να μειώνεται κατά 10% για παράδειγμα η χρηματοδότησή σας. Να υπάρχουν αυτές οι συνέπειες γιατί αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Ε, όταν θεωρούμε πως δεν μπορεί να δοθεί η απαλλαγή. Την επόμενη λοιπόν περίοδο πιστεύω πως θα πρέπει να δράσουμε με τον τρόπο αυτό. Θα πρέπει να παρέμβουμε, θα πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη αξιολόγηση, να δούμε ποιο είναι το άλλο το υπόλοιπο πρόγραμμα που μας μένει μπροστά μας, τι λένε τα άλλα όργανα και να μπορέσουμε να μπούμε και στο κομμάτι του πολιτικού σχεδιασμού για τα διάφορα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται εδώ. Και τι σημαίνει σε περίπτωση που έχουμε συνδιαχείριση, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί πάντοτε. Να πω και ένα τελευταίο, χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Την τελευταία περίοδο θελήσαμε μέγιστη διαφάνεια για να αποφύγουμε την απάτη και τις πολιτικές επιρροές στα κράτη-μέλη ή την επιρροή τρίτων χωρών. Θα πρέπει όμως να δούμε τι γίνεται, πώς επηρεάζουν τις χώρες μας, η Ρωσία, η Κίνα, που θέλουν ακόμα και εκλογικά αποτελέσματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χειραγωγήσουν. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα ξεκάθαρο ε, ρόλο να παίξει και σας ευχαριστώ που δώσετε χρόνο να σας παρουσιάσω την εκθέση. Ähm, ευχαριστώ. Να ζητήσω συγγνώμη για τη θερμοκρασία της αίθουσας. Ε, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει γιατί κάνει τόσο κρύο, ο τεχνικός ε, λείπει. Πραγματικά κάνει πάρα πολύ κρύο εδώ πάνω. Δεν ξέρω τι γίνεται και στις καμπίνες, ζητώ συγγνώμη. Θα, θα διέκοπτα τη συνεδρίαση, αλλά έχουμε τόσο πολλά πράγματα στην μέση διάταξη που δεν ε, γίνεται. Ναι, ναι, το απόγευμα να απαντάει σε σχόλιο εκτός μικροφώνου η πρόεδρος. Κυρία Μπουσκές για την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Σκεντόφσκι. Σωστά η η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στο θέμα της λογοδοσίας και του μηχανισμού ελέγχου. Όλες οι ακροάσεις που γίνονται εδώ με γενικούς διευθυντές, με επιτρόπους, με το Γενικό Γραμματέα σήμερα είναι στιγμές κλειδιά για εμάς για να βελτιώσουμε την δημοσιονομική διαχείριση για να δούμε ποια είναι τα βασικά σημεία και τα αποτελέσματα του κοινοτικού προπολογισμού. εδώ. Χωρίς να μπω σε λεπτομερίες θα ήθελα να επισημάνω ότι η απόδοση και οι εκθέσεις ε, που αφορούν αυτό το θέμα πλέον αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία και βελτιωνόμαστε ως ε, προς αυτό. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα στιβαρό πλαίσιο απόδοση, αλλά ακούγοντα και τις προτάσεις σας η Κομισιόν πρότεινε να υπάρξει μια ευθυγράμμιση του πλαισίου αυτού στον νέο κανονισμό επίσης ε, στο νέο ΠΔΠ, επίσης στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται αρχή απαλλαγής για την ε, διαδικασία αυτή και όλες τις πληροφορίες που είναι σημαντικές και για τους ε, πολίτες. Γιατί τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξηγούμε το πώς εξοδεύουμε τον προϋπολογισμό αλλά και ποια αποτελέσματα έχουμε. Η Κομισιόν παίρνει πολύ στα σοβαρά την ε, διαδικασία της απαλλαγής και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις της ε, διαδικασίας. Και μετά την απαλλαγή οι υπηρεσίες της Κομισιόν αναλύουν όλες τις συστάσεις ε, και προετοιμάζουμε μια έκθεση για εσάς, για όλες τις δράσεις που έχουμε αναλάβει ή θα αναλάβουμε στο μέλλον. Το ίδιο έχει γίνει και εδώ για την πρόταση του επόμενου ΠΔΠ. Θα ήθελα καταλήγοντας να επιβεβαιώσω ότι η προσπάθεια αυτή αποδίδει καρπούς. Στην έκθεση αναφέρεται ότι είναι καλύτερη η δημοσιονομική διαχείριση της Ένωσης από ό,τι στο παρελθόν. Ο Επίτροπος Έτιγκερ είπε ότι η διαδικασία της απαλλαγή διδάσκεται από το παρελθόν και από τον τρέχοντα μηχανισμό. Και θα θέλαμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την δημοσιονομική διαχείριση και ακριβώς ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να σας πω πως η προθεσμία είναι 4 Δεκεμβρίου 2 η ώρα και μετά θα μας απασχολήσει ξανά αυτό το θέμα με το νέο έτος και θα ασχοληθεί η ΑΦΚΟ στις 22 Ιανουαρίου. Περνάμε σημείο 16. Την έκθεση ε, για την καταπολέμηση της απάτης ε, και την προστασία των ομιλών συμφερόντων της Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκο. Έχετε το λόγο. Να σας πω λοιπόν για το κρύο πως αυτό σημαίνει ότι ενεργειακά είμαστε αποδοτικοί. Μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος. Αν κρυώνουμε φταίνει πράσινη. Είμαι σίγουρος. Έτσι έχει κατάσταση, κυρία Πρόεδρε. Έχετε το φάκελο μπροστά σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο φάκελος αυτός, δεν θα πω ότι είναι σημαντικός. Έχετε διαβάσει, είναι όλα τα στατιστικά δεδομένα σε σχέση με το θέμα αυτό. Αυτό το οποίο επιθυμώ να πω στα γρήγορα είναι πως υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα ο Γενικός Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική αυτή η εισαγγελία και να δώσει τη μάχη με αποτελεσματικό τρόπο ε, κατά της απάτης και άλλων σχετικών. Και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, να πιέσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνεργασία. Δεύτερον, ψηφιοποίηση. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να πατάξουμε την απάτη, αλλά θα πρέπει να προλάβουμε και την απάτη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μπορούμε να πούμε ότι ότι έχουμε εξοικονομήσει ε, χρήματα με συγχωρείτε, και προσπάθειες ε, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε και να μην χρειάζεται απλώς να διώκουμε την απάτη. Τώρα με την πρόοδο της τεχνολογίας είναι πολύ εύκολο. Ψηφιοποίηση λοιπόν για όλες τις διαδικασίες της εφαρμογής του προϋπολογισμού και των έργων. Ξεκινάμε λοιπόν με την προκήρυξη, με την εφαρμογή, με το διαγωνισμό, με τις πληρωμές. Όλα αυτά σε ένα έργο θα πρέπει να γίνονται σε μια ψηφιοποιημένη πλατφόρμα. Κάποιο κράτη-μέλη το κάνουν ήδη, είναι πολύ λίγα. Και προτείνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθεί ένα πλαίσιο έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό και να το εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη. Όντως υπάρχουν προβλήματα, όντως υπάρχουν διάφορα θέματα με τις ε, οδηγίες για τις κρατικές πριμήθειες, όμως θα τα καταφέρουμε και πιστεύω ότι θα εξοικονομήσουμε και πολλά κονδύλια. Έτσι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τους ε, σκιώδεις. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης ηγητής για αυτό το θέμα. Ο Μπένιντεκ Διάβορ είναι. Μου ζήτησε όμως να μεταφέρω τα όσα έχει να πει. Ευχαριστή τον κύριο Μαρινέσκου για την έκθεση. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ετήσια έκθεση αυτή αλλάζει από το ένα έτος στο άλλο και υπάρχει ακριβώς ε, η ετήσια ανασκόπηση της ε, κατάστασης για να υπάρξει ακριβώς η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Και το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Η έκθεση αυτή λοιπόν, όπως ε, μας λέει ο κ. Γιώβαρα εδώ πέρα, ε, διαφέρει στο εξής, ότι τώρα έχουμε το τελευταίο έτος ε, της θητείας μας και κάνουμε έναν απολογισμό των όσων συνέβησαν τα τελευταία πέντε χρόνια για να δούμε ποια είναι τα πιο προβληματικά σημεία οπωσδήποτε. Σύμφωνα με τον συνάδελφό μου υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις στο πλαίσιο της, ε, του κανονισμού Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε την οδηγία περί ε, καταγγελόντων, αλλά ο Μπέντικτ Γιάβορ θεωρεί ότι εδώ πέρα έχουμε έναν ε, τομέα ο οποίος έχει απαξιωθεί ε, και μιλάει συγκεκριμένα για την καταπολέμηση της διαφοράς έχει εφετηθεί ένα πακέτο κατά της ε, διαφθοράς και ο Μπένεντικτ θεωρεί ότι από το 2011 η κατάσταση δεν έχει αλλάξει πολύ. Έχουμε δηλαδή την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον Κρεκο, που είναι πολύ περιορισμένη. Η έκθεση κατά της ε, διαφθοράς εγκαταλείπεται η διαφορά ανθίζει και η διασυνοριακή εγκληματικότητα και η απάτη του ΦΠΑ εξακολουθούν να ανθούν και τα κονδύλια τα οποία μοιράζονται στα κράτη-μέλη συχνά συνδέονται με διαφορά εκεί και καταλήγει ο συνάδελφος ε, κύριε Πρόεδρε στο ότι πιθανώς ε, θα υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες για να μπορέσει να αναλύσει καλύτερα την κατάσταση με στόχο τελικά το επόμενο κοινοβούλιο, η επόμενη θητεία μέσω της έκθεσης αυτής να έχει μια εποπτεία των συστάσεων αυτών. Υπό αυτήν την έννοια ο Μπένεντικτ Γιάβορ θα υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες ε, για να ενισχύσει το κείμενο στο θέμα του Όλαφ, ε, στο θέμα του ΦΠΑ σε συνεργασία με εσά και τους άλλους ε, σκιώδεις Αυτά θα σας έλεγε ο Μπενετιά αν ήταν εδώ. Σας ευχαριστώ. Να ήθελα και εγώ να πω κάτι για τις τροπολογίες που θα υποβάλω εγώ. Βεβαίως ε, έχουμε το θέμα του Όλαφ και του πληροφοριακού συστήματος του το οποίο δεν λειτουργεί και έχουμε εδώ πέρα πραγματικά την αχίλιο πτέρνα του Όλαφ γιατί ε, μπορεί να εξαφανίζονται ολόκληρες περιπτώσεις ε, και υποθέσεις από εκεί μέσα. Οπότε θα το καλύψω αυτό με κάποιες τροπολογίες. Και βέβαια αν δούμε και την έκθεση του Όλαφ βλέπουμε ότι υπάρχουν ασυνέπειες στην ορολογία και δεν υπάρχει συγκρισιμότητα σε βάθος χρόνου. Και θα ήθελα να δούμε και κάποια πράγματα όσον αφορά τις περιπτώσεις απάτης και την επεξεργασία τους. Γνωρίζω ήδη ότι η έκθεση αυτή βασίζεται σε ένα έγγραφο της ε, Κομισιόν και βεβαίως ε, χρειαζόμαστε ακριβώς ε, το θέμα αυτό της ε, καταπολέμησης αβάτης. Τα θέμα των δημοσίων προμηθειών είναι πάντα ένα θέμα που μας απασχολεί. Πρέπει να δούμε δηλαδή το τι θα γίνει με τις απλές τακτικές διαδικασίες προμηθειών, πώς θα τις παρακολουθούμε προσεκτικότερα στα κράτη-μέλη, γιατί οι περιπτώσεις απάτης ε, δεν αφορούν πλέον κάποια πλαστογραφημένα έγγραφα, είναι πολύ πιο έξυπνες. Χρησιμοποιούν τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στείνονται διαγωνισμοί, παραδείγματο χάρη, ε, που θα έπρεπε να είναι αντικείμενο ανοιχτού ανταγωνισμού. Το κείμενο λοιπόν είναι καλό και καλό θα είναι να το βελτιώσουμε. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο τον λόγο. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στην κυρία Χόφμαν από τον Όλαφ. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Μαρινέσκου για την πολύ καλή αυτή έκθεση. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά. Χαιρόμαστε που ο εισηγητής αναγνωρίζει ε, θετικά τις διάφορες πρωτοβουλίες του 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς. Στην εκθεσή σας ε, υπογραμμίζετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Επιτροπή, η DG Olaf και η DG Justice ε, βρισκόμαστε σε εντατικές προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να τεθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε λειτουργία στα τέλη του 2020. Οπότε καλωσορίζουμε οποιαδήποτε υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το μέτωπο. Επίσης αναφέρατε το σύστημα πρώιμης ανείχνευσης και αποκλεισμού που λειτουργεί καλά και το άλλο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της απάτης με στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από δική μας άποψη, στην Κομισιόν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της απάτης και χέρμα που συμφωνείτε κι εσείς. Συνολικά έχω να κάνω μια παρατήρηση που δεν αναφέρθηκε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες που ο κύριος Μαρινέσκου, κύριε Μαρινέσκου που συμπεριλάβατε κάποια σημαντικά στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν. Αναγνωρίζετε το ότι ο αριθμός των εντοπισμών μπορεί να οφείλεται στις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη και όχι στο πόσα περιστατικά υπάρχουν πραγματικά. Αυτή τη συζήτηση έχει γίνει εδώ και καιρό, γίνεται εδώ και καιρό στην Επιτροπή Κόντο. Ε, θέλει κάποια ισορροπία, δύο στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οπότε χαιρόμαστε που στην έκθεση αυτή αναγνωρίζεται ρητά αυτή τη δυνατότητα ανείχνευσης των κρατών μελών. Εάν ένα κράτος μέλος δηλαδή ε, αναφέρει πολλές περιπτώσεις ε, απάτης ε, και παρατυπιών. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι ικανότητες ανείχνευσης είναι πολύ καλές στο κράτος μάλλον αυτό. Κάτι άλλο που αναφέρατε στις παρατηρήσεις σας εμείς στην Επιτροπή είμαστε υπέρα της ενισχυμένης ψηφιοποίησης όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Τις προτάσεις λοιπόν τις λαμβάνουμε υπόψη Έχουμε το πλαίσιο της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις ε, και συνεργαζόμαστε με την DigiGrow η οποία συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η ψηφιοποίηση και συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τις απάτε στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Σημειώνω τα όσα είπε ο κ. Στάς σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τη συζήτηση αυτή την έχουμε ξανακάνει το γιατί η Κομισιόν ε, δεν ε, ε, εκδίδει πιο συχνά εκθέσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για την καταπολέμηση αυτού του φλέγοντος ζητήματος. Συμφωνώ μαζί σα. Πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εξετάστηκε μάλλον στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εκεί είδαμε κάποια πρόοδο. Συμφωνούν και τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη επιμονή και να συνεργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη. Και πρέπει να δείξουμε και κάποια σκληρότητα με τα κράτη-μέλη. Έχετε δίκιο. Για την Όλαφ, ε, η καταπολέμηση της διαφθοράς ε, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Συχνά μάλιστα παρευρισκόμαστε σε εκδηλώσεις μαζί με τα κράτη-μέλη για να προωθήσουμε την καλύτερη, την ενισχυμένη ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Γκρέσλε και τις παρατηρήσεις τη, Αναφέρατε το σύστημα μας ε, πληροφορικής, στο OCM, όπως ονομάζεται, που είναι το νέο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων στην Όλαφ. Δεν είναι μυστικό ότι είχαμε κάποια προβλήματα με αυτό το νέο σύστημα. Ο νέος κοινικός μας διευθυντής, ο κ. Σιτάλα, νομίζω και εδώ στην Επιτροπή σας έχει αναγνωρίσει ήδη ότι έχουν γίνει εντατικέ ε, ενδελεχείς προσπάθειες για βελτίωση της λειτουργίας και υπάρχουν και βελτιώσεις ήδη ορατές. τα ανώτατα στελέχη το παρακολουθούν στενά. Αλλά είμαι βέβαιο ότι κυρία Γκρέσλε, κυρία Γκρέσλε, όταν θα υποβάλλετε εσεί τροπολογίε, θα τι δούμε και εμεί και να είστε βέβαιοι ότι και ο δικό μα Γενικό Διευθυντή παρακολουθεί στενά το ζήτημα. Επίσης αναφέρατε κάποια θέματα συνέχεια ε, στην ορολογία, αλλά είπατε επίσης ότι η έκθεση Όλαφ και η έκθεση ΠΥΦ βασίζονται σε διαφορετικές μετρήσεις. Η έκθεση της Όλαφ βασίζεται στο δικό μας σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και στις υποθέσεις με τις οποίες ασχολούμαστε εμείς στην Όλαφ. Η έκθεση ΠΥΦ ασχολείται με την ανάλυση των εκθέσεων των κρατών μελών για παρατυπίες ε, ε, που οφείλονται σε απάτη και που δεν οφείλονται σε απάτε. Ε, ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Απλά ήθελα να επισημάνω αυτέ τι δύο διαφορετικέ προσεγγίσεις που θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε και να λάβουμε υπόψη. Συνολικά είμαστε ικανοποιημένοι με την εκθέση αυτή ε, και με το γεγονό ότι εξετάζει το θέμα κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο. Προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία μαζί σα και με τον εισηγητή και περιμένουμε και τι τροπολογίε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χόφμαν. Ήθελα να διευκρινίσω ότι η κριτική μου για τα θέματα ορολογίας δεν αφορούσαν την Όλαφ και το ΠΙΦ, αλλά την Όλαφ μόνο. Ε, δεν ξέρει κανεί όταν κοιτάει κάποιε λέξει αν πρόκειται για τα ίδια πράγματα. Investigations closed και concluded είναι το ίδιο, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Πρέπει να δούμε, έχετε και στη βάση δεδομένων ε, πόσες ε, εταιρείε υπάρχουν εκεί, ε, πόσες... maybe... Δεν ξέρω, αλλά ίσως ο κύριος Μίσλικ που είναι αρμόδιος στην Όλαφ μπορεί να γνωρίζει παραπάνω η DG Budget είναι ε, η Γενική Διεύθυνση που είναι υπεύθυνη. Κάναμε μια συνάντηση λοιπόν πρόσφατα μαζί τους και στο πάνελ μας είπαν πως μέχρι στιγμής έχουν οκτώ υποθέσεις τις οποίες έχουν λάβει και έξι ε, ακόμα είναι ανοιχτέ. Είναι πάντως μια νέα διαδικασία και η συνεργασία αυτή τη στιγμή πάει καλά με την Γενική Διεύθυνση Budget αλλά λόγω των επιπέδων της χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε. Ξέρετε τι έγινε στο παρελθόν. Είχαμε ένα ευρωπαϊκό εσωτερικό σύστημα και το ΔΕΚ θεώρησε πως αυτό παραβιάσει το δικαίωμα ακρόασης. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε το πάνελ με την προεδρία του κυρίου Πανέρα για να εξασφαλίζεται πως όλα γίνονται σύνομα. Είναι μια σχετικά νέα διαδικασία ε, και εκεί έχουν κάποιες ανοιχτές υποθέσεις που είναι σημαντικές, αλλά η συνεργασία πάει πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Φτάσαμε στο τέλος. Εισηγητή έχει το λόγο για να κλείσουμε. Παρακαλώ. yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που κάνατε. Νέο κεφάλαιο, λεφτό, νέο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, μάχη κατά της διαφθοράς. Αυτό θα έπρεπε να εισαχθεί μέσω των τροπολογιών σας, τις οποίες περιμένω και περιμένω και τις βελτιώσεις που θα προτείνετε και ελπίζω πως η έκθεση θα είναι καλή. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για τροπολογίες 26 Νοεμβρίου 2 η ώρα και στις 13 ε, Δεκεμβρίου θα μας απασχολήσει το θέμα στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης. Χωρί μικρόφωνο η πρόεδρο. Α, ναι, ναι, συγγνώμη. Ο εισηγητή απουσιώζει, οπότε θα πω εγώ κάτι πράγματα. Να υπενθυμίσω ότι Έχουμε εδώ πέρα μια γνωμοδότηση για την σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Το θέμα λοιπόν εδώ πέρα είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, το ESM το οποίο δημιουργήθηκε υπό συνθήκες κρίσης, να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο για να διασφαλίσουμε την σταθερότητα της Ευρωζώνης ο μηχανισμός σταθερότητας μερίθηκε το 2012 ως ε, διακυβερνητική συνθήκη και ακριβώς ένα χρόνο μετά ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεταφερθεί ο μηχανισμός στο κοινοτικό δίκαιο. Κάτι το οποίο τελικά συνέβη η Κομισιόν ε, ε, ζήτησε κάτι τέτοιο. Οπότε Γαλλία και Γερμανία έκαναν μια κοινή δήλωση και γι' αυτό ακριβώς ε, έχουμε και τη σημερινή μας γνωμοδότηση. Ο συγγητή χαιρετίζει την πρόταση αυτή η οποία βεβαίως καταφέρνει να ανταποκριθεί σε ένα πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο θα ενισχυθεί και η λογοδοσία. Προτείνει ο συγητής ε, να υπάρξει αυξημένος ρόλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και το ταμείο αυτό να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με την διαδικασία της απαλλαγής. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει έναν ρόλο στον ορισμό του Διευθυντή και θα γράφετε και μια, θα υποβάλλετε μια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν. Θα ήθελα, δεν έχεις δει κάποιο τον λόγο, οπότε θα δώσω τον λόγο στον κύριο Έγγελεν. Α, συγγνώμη, Κρόμποκ της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΦΙΝ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του εισηγητή για την πρόταση από το Δεκέμβριο του 2018 και συντάσσεται απόλυπα ε, με τα όσα έχει στην γνωμοδότηση όπου ζητά να υπάρχει ε, μια κοινοτική εντολή στη βάση όλων των προτάσεων που θα κάνουμε στα πλαίσια της αναθεώρησης της ε, ΟΝΕ με τρόπο που θα έχουμε μεγαλύτερη δημοκρατική επιλεξιμότητα. Για το σχέδιο γνωμοδότησης έχουμε συγκεκριμένα σχόλια Καταρχήν, θα ήταν βιώσιμο να έχουμε καλύτερη άρθρωση των σχετικό ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου ε, στα σημεία 6, 8 και 9 του, του σχεδίου γνωμοδότησης. Καταγράφουμε εδώ πως το, ε, ε, η αιτιολογική σκέψη 64 της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής αναφέρεται στο ότι το ελεγκτικό συνεδρίο μπορεί να ασκεί πλήρω τις αρμοδιότητές του και μπορούμε να δούμε μαζί με εσά και τα κράτη-μέλη πώς μπορεί ο ρόλος αυτός του ελεγκτικού συνεδρίου να ε, διατυπώνεται καλύτερα στα πλαίσια της πρότασής μας. Τώρα, για την αναφορά που γίνεται στην ε, αντικατάσταση, στην υποκατάσταση των εξωτερικών ε, ελεγκτών που έχουμε στην τρέχουσα συνθήκη για την ΟΝΕ, πιστεύουμε πως όλα αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν δεδομένου του ότι η ΟΝΕ είναι μια χρηματοδοτική πλατφόρμα που ε, λειτουργεί στι διεθνεί αγορές και θα πρέπει να πιστοποιούνται επαρκώς οι λογαριασμοί του έτσι ώστε οι επενδυτές να αισθάνονται πως μπορούν άνετα να επενδύσουν στα ομόλογα που εκδίδει. Και να σα υπενθυμίσω πως αυτό δεν είναι ασυνήθιστο γιατί έχουμε κάτι αντίστοιχο στη συνθήκη για την ΕΚΤ και για τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των Κρατών Μελών. Για το ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαδικασία του διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή, άρθρο 7 ε, του σχεδίου καταστατικού που ακολουθεί την νομοθετική μας πρόταση, όπου το Συμβούλιο θα πρέπει να διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή να παίξει έναν ενεργό ρόλο. Και για τη λογοδεσία, 10, 11 και 12 σημεία της γνωμοδότησης καταγράφουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βασίσει τις ε, ε, σχετικές διατυπώσεις ε, στα πλαίσια των διεθνών προτύπων που έχουμε σε άλλη δευτερεύουσα νομοθεσία, για παράδειγμα το Single Resolution Board και τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και έχει προβλέψει αυτή η δυνατότητα να υπάρχει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει απόρριτες ακροάσεις, έτσι ώστε να ασκήσει το ρόλο του που είναι αυτός του επόπτη. Ευχαριστώ. Οπότε φτάνουμε στις τροπολογίες. 21 Νοεμβρίου, αύριο δηλαδή, στις 2 η ώρα είναι η προθεσμία και στις 13 Δεκεμβρίου θα μας απασχολήσει ξανά το θέμα. Άρα τελειώσαμε αυτό το θέμα της μέσης διάταξης. Σας ευχαριστώ και τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί συνεχίζουμε. ωραία, ωραία.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 από τη DG Budget. Ο κ. Κόπμαν. Κανείς δεν είναι. Ε, από την DG Ample επίσης δεν βλέπω κανέναν. Ε, είμαστε αναγκασμένοι άρα να διακόψουμε μέχρι αξιότιμοι κύριοι και κυρίες ε, ελπίζω να, να ειδοποιηθούν και να έρθουν. Περιμένουμε να έρθουν. Ε, είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς τον χρόνο. Συνήθως είναι το αντίθετο πρόβλημα. Καθυστερούμε. Ε, μόλις έρθουν λοιπόν οι αρμόδιοι θα συνεχίσουμε αμέσω με το θέμα αυτό των αντικρώμενων συμφερόντων και αυτό το οποίο συζητήσαμε με τον Επίτροπο το πώς δηλαδή η Κομισιόν θα εφαρμόσει το άρθρο 61. Solange bis die Διακόπτεται λοιπόν η συνεδρίαση. Ja, wir nehmen unsere Beratungen nach kurzer Unterbrechung wieder auf. Und Gegenstand. Συνεχίζουμε μετά από το διάλειμμα. Χαιρετίζω την Γενική Διεύθυνση και τον νέο Γενικό Διευθυντή του Προπολογισμού, κύριε Κόκμαν. Δεν σας είχαμε ξαναδεί. Έχουμε τον κύριο Ζέμπερτ από τη Γενική Διεύθυνση Ζέμπερτ και η κυρία Μπόχημαν δεν έχει έρθει. Ελπίζω να έρθει κάποια στιγμή. Και Α, πιαν, πιαν, τη, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας εκπροσωπεί. Ρέγγιο, ναι, μάλιστα. Και μας λείπει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως ε, εξής. Άρθρο 61. η Δημοσιονομική φορείς στο πλαίσιο του ορισμού του άρθρου 4 περιλαμβανομένων των εθνικών αρχών σε οποιοδήποτε επίπεδο που εμπλέκονται στην εκτέλεση του προπολογισμού σε άμεση και έμεση και κοινή διαχείριση που ασκούν έλεγχο ή εσωτερικό έλεγχο δεν θα αναλάβουν δράση η οποία θα φέρνει τα συμφέροντά τους ε, σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Ένωσης. Επίσης ε, θα λάβουν μέτρα για να μην προκύψει σύγκρουση συμφερόντων εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους ε, και καταστάσεις οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ως αντικρόμενα συμφέροντα. Εδάφιο 2. Όπου υπάρχει τέτοιος κίνδυνος ε, με μέλος του προσωπικού της Εθνικής Αρχής, ε, τον λόγο άτομο θα παραπέμψει το ζήτημα στους ανωτέρους του. Στην ε, περίπτωση αυτή θα αναπαινθεί το ζήτημα στον ιεραρχικά ανώτερο, ο οποίος θα επιβεβαιώσει γραπτός εάν υπάρχει η περίπτωση αντικρόμου σφαιρότων. Στην περίπτωση που ισχύει αυτό, θα διασφαλιστεί το ότι το εν λόγω άτομο θα σταματήσει να εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό. Και η αρμόδια εθνική αρχή θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε άλλη ε, δράση θα αναλαμβάνεται συμφώνως ε, προς ε, το ισχύον δικαίωμα. Τρίτον, υπάρχει υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα στην περίπτωση στην οποία δεν είναι δυνατή η άσκηση αντικειμενικής λειτουργίας για λόγους οικογενειακούς ε, ή πολιτικών ή άλλων δεσμών ή οποιοδήποτε άλλου άμεσου ή έμεσου συμφέροντος. Αυτά λέει το άρθρο 61. Και το καινούργιο βεβαίως είναι η συμπερίληψη των εθνικών αρχών και εθνικών πολιτικών. Και εμείς ανησυχούμε γιατί βλέπουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει μια κατάσταση όπου ε, πρέπει, θα έπρεπε να εφαρμοστεί και να ισχύσει κατεπηγόντως αυτό το άρθρο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Ε, έχουμε κάποια παραδείγματα εδώ κατά νου. Είναι μια πρόκληση λοιπόν ε, που ξεπερνάει θα έλεγα τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα σε μια κρυα αίθουσα και το ερώτημα είναι ποιος από τους κυρίους θέλει να λάβει πρώτος τον λόγο. Εσείς κύριε Κούκμαν παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τους κανόνες και το νέο οικονομικό κανονισμό για τα σύγκρουση συμφορώντων. Έχω συμφωνήσει με τους συναδελφούς μου να σας κάνουμε μια παρουσίαση της γενικής εικόνας του πώς το βλέπουμε εμείς τις ευθύνες των εθνικών παραγόντων και της Επιτροπής σύμφωνα με την Επιτροπή. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν ε, βήμα-βήμα την παρουσίαση όπου διατυπώνονται οι απόψεις μας και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον προϋπάρχοντα οικονομικό κανονισμό που υπήρχε πριν από τις 4 Αυγούστου φέτος γιατί προφανώς ε, διάφορες υποθέσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή και στις οποίες νομίζω αναφερθήκατε ε, εξαρτώνται από αυτόν. Όπως βλέπετε, ο οικονομικός κανονισμός του 2012 δεν αφορούσε ρητά την επιμερισμένη διαχείριση όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Ωστόσο, και αυτό είναι σημαντικό να το σημειώνουμε, ανέφερε προφανώς ότι τα κράτη-μέλη έπρεπε να διασφαλίζουν αποτελεσματικούς εσωτερικούς ελέγχους και τα σχετικά συστήματα που θα έπρεπε να μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς και τις περιπτώσεις πιθανών ε, συγκρούσεων συμφερόντων και να τις αποφεύγουν. Θέλω να επισημάνω τα άρθρα 32, 3 και 59, 4 λοιπόν του οικονομικού κανονισμού του 2012. Το άρθρο 24 της οδηγίας 2014-24 επίσης ε, επιτρέπει την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων γιατί αυτό αυτή η οδηγία είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η οδηγία αυτή καλύπτει επίσης και τις περιπτώσεις ε, υποψίας ε, σύγκρουσης συμφερόντων και αναφέρεται και σε άμεσα και σε έμεσα σύγκρουση συμφερόντων περισσότερα συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους κανόνες επιμερισμένης διαχείρισης υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ειδικότερα στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, για να σας δώσω κάποια παραδείγματα, το άρθρο 5.3, το 34.3 και το 38.5 ε, αφορούν αυτό το θέμα της επιμερισμένης διαχείρισης. Αν δούμε την αγροτική πολιτική, να παραθέσω εκεί την κατεξοδότηση ε, κατεξοδότηση πράξη την 907-2014. Τι λέω εδώ λοιπόν ότι όσον αφορά την κατάσταση πριν από τις 2 Αυγούστου 2018 είχαμε ήδη διάφορους κανόνες και ο κανονισμός που έχει τεθεί τώρα σε ισχύ βασίζεται στους κανόνες αυτούς και τους επεκτείνει, τους κωδικοποιεί ουσιαστικά σε κεντρικούς κανόνες που αφορούν ε, την ε, οικονομική διαχείριση γενικότερα της Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, το αναφέρατε, οπότε δεν θα μακρηγορήσω από αυτού, οι κανόνες ε, τέθηκαν σε ισχύ στις 2 Αυγούστου για, τη, ε, επιχειρησιακά, για τις επιχειρησιακές πιστώσεις και 1 Ιανουαρίου του 2019 όσον αφορά τα διοικητικά κονδυλία. Αναφερθήκατε στο άρθρο 61 που πράγματι ε, θεσπίζει τους βασικούς κανόνες ε, για τη σύγκρουση συμφερόντων. Να σας τονίσω τα νέα ε, σημεία εδώ που βασίζονται σε αυτά που ανέφερα. Στον ορισμό λοιπόν τη σύγκρουση συμφερόντων, τι νέο υπάρχει και το υπογραμμίζω η αναφορά στα έμεσα προσωπικά συμφέροντα. Αυτά τώρα καλύπτονται ρητά. Στο ποια υπόκεινται σε αυτό το ε, κανονισμό οι φορείς είναι όλες οι εθνικές αρχές οποιοδήποτε επίπεδου που καλύπτονται από αυτό το κανονισμό και η επιμερισμένη διαχείριση επίσης καλύπτεται ρητά από τον οικονομικό κανονισμό. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη οπωσδήποτε ότι οι ρητές αναφορές ε, ε, στον κανονισμό θα ισχύουν υπέρ οποιοδήποτε κανόνων υπήρχαν. Και εδώ καθορίζεται πολύ σαφώς σε ποιον αφορούν οι κανόνε αυτοί. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι προβλέπονται δράσεις εδώ υποχρεωτικές για την αποφύγη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που οδηγούν σε παρατυπίες όσον αφορά τη διαχείριση κονδυλίων. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο πρώτο άρθρο. στο πρώτο κομμάτι αυτού του άρθρου και αυτό που λέει εδώ είναι κάτι νέο. Λέει ότι στις περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν ε, ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Οι φορείς ε, απαιτείται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί να λάβουν χώρα. Αυτό προέρχεται από τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων ότι πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων που αντικειμενικά μπορεί να θεωρηθούν σύγκρουση συμφερόντων. Εδώ δηλαδή έχουμε μια νέα ρητή απέτηση για όλους τους φορείς να αναλαμβάνουν δράση ούτω ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπόθεση ότι υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Το νέο σε σχέση με τις δημοσίες συμβάσεις εδώ είναι η λέξη αντικειμενικά. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή την εικόνα που δίδεται ε, της σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπλέον τώρα, όσον αφορά τις υποχρεώσεις και εδώ νομίζω η πρόεδρος ε, το ανέφερε. Εάν ε, ένα μέλος του προσωπικού μιας εθνικής αρχής ε, αν σε αυτόν εφαρμόζεται κάποιο σύνολο από αυτόν τον κανόνων όπως έχει κωδικοποιηθεί πολύ σωστά, θα ισχύουν γι' αυτόν αυτοί οι κανόνες. Για να συνοψίσω τώρα τι νέο έχουμε στο άρθρο 61, την αναδιατύπωση του ορισμού της σύγκρουσης συμφερόντων. Τώρα ρητά αναφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμεσο προσωπικό συμφέρον. Δεύτερον, ότι οι καταστάσεις, οι περιπτώσεις που καλύπτονται είναι πιο πολύ αριθμές, έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή, διότι καταστάσεις που μπορεί κανείς αντικειμενικά να θεωρήσει σύγκρουση συμφερόντων καλύπτονται επίσης ρητά και επίση, όσον αφορά τον τύπο των δράσεων, έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή. Όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση, και τη ρητή αναφορά ότι οι εθνικέ αρχές οποιοδήποτε επίπεδου πρέπει να αποφεύγουν και να διαχειρίζονται αυτές τις συγκρούσεις συμφερόντων. Εδώ πιστεύω συνοψίζεται λοιπόν πολύ σαφώς η εξέλιξη της Ευρωπαϊκή Δημοθεσία από αυτήν την ε, άποψη που έχει ψηφιστεί και εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι ύψη τη σημασία φυσικά για το έργο που καλείται να επιτελέσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Δεδομένου ότι πρόκειται για κάτι καινούργιο, θέλω να εστιάσουμε λίγο στην ε, ε, εικόνα αυτή ε, μια σύγκρουση συμφερόντων, στην υποτιθέμενη σύγκρουση συμφερόντων, όπως είπα, ευθυγραμμίζεται με την οδηγία για τις δημοσίες συμβάσεις και έχει προσθεθεί αυτό η, έννοια της αντικειμενικής επαλήθευσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τέτοιου στοιχείου αντικειμενικά επαλήθευση μου κάποια σχέση μεταξύ του εν λόγω ατόμου και φορέων όπου έχουν αναλαβεί την ευθύνη ε, για οικονομικές αποφάσεις, για αποφάσεις οικονομικής διαχείρισης. Αυτές οι διευκρινήσεις πιστεύω είναι σημαντικές. Μας βοηθούν να ανοιχνεύσουμε οποιασδήποτε περαιτέρω ε, υποθέσεις. Παρομοίως η έννοια ότι υπάρχει ε, ε, οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμεσο προσωπικό συμφέρον το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί ε, τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό είναι ευρύτερο από την παλιά διατύπωση στο άρθρο 57 του προηγούμενου οικονομικού κανονισμού, του κανονισμού για τις δημοσιονομικούς κανόνες. που αναφερόταν απλά σε δικαιούχου. Είναι σημαντικό για όσου έχουν κοιτάξει τον δημοσιονομικό αυτό κανονισμό να λάβουν υπόψη το γεγονό ότι οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιες ε, ε, διαφορές ε, απαριθμώνται επακριβώς αναφέρονται σε οικογένεια, συναισθηματική ζωή, πολιτική ζωή, οικονομικά συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο. Απαριθμεί δηλαδή το άρθρο με μεγάλη ακρίβεια το πρόβλημα αυτό όσον αφορά τα άτομα τα οποία αφορά η επιμερισμένη διαχείριση και εκεί είναι απολύτως σαφές ότι περιλαμβάνονται οι εθνικές, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές προσωπικό και μέλη του προσωπικού των αρχών αυτών και ε, κυβερνητικά στελέχη. Αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναθεώρηση του ε, κανονισμού για τις νομικούς κανόνες ε, με αυτή τη συγκεκριμένη διατύπωση που σχετίζεται με τις εθνικές αρχές που προσθέθηκε κατά τους τριλόγους μετά από αίτημα νομίζω της Επιτροπής αυτής εδώ. Και συμπεριλήφθηκε και σαφής αναφορά και στα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχει καθοριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογή. Για να κλείσω τώρα. Είναι σημαντικό αφού έχουν διευκρινιστεί όλα αυτά να είμαστε ακριβείς όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Κομισιόν για την αντιμετώπιση τέτοιων πιθανών περιπτώσεων. Τα κράτη-μέλη λοιπόν υποχρεούνται να καθιερώσουν εσωτερικά συστήματα ελέγχου σχεδιασμένα ώστε να διασφαλίζουν αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων ή τηρητή διαχείριση τέτοιων συγκρούσεων συμφερόντων. Υποχρεούνται επίση τα κράτη-μέλη ε, τη σωστή στελέχωση αυτών των συστημάτων και τη σωστή του λειτουργία. Δεύτερον, πρέπει να καθιερώνουν προληπτικά μέτρα, όπω για παράδειγμα τα συστήματα δηλώσεων που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη όσον αφορά την απουσία ε, συγκρούσεων συμφερόντων, ε, ε, δημοσιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, όπω απαιτεί και Κομισιόν. Τρίτον, πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα θα έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ούτω ώστε κάθε φορά που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων να υπάρχουν και να υλοποιούνται και τα απαραίτητα μέτρα, ε, διορθωτικά μέτρα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν βάσει των κανόνων έχουν αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά θέλω να το πω τώρα σαφώς. Δεν, δεν είναι ότι η Κομισιόν δεν έχει καμία υποχρέωση. Αντιθέτω, απαιτείται από αυτήν να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εθνικών συστημάτων με τις ευρωπαϊκές απαιτήσει. Εμείς πραγματοποιούμε ελέγχους στα εσωτερικά συστήματα ελέγχου των κρατών μελών βάσει επικινδυνότητας. Αυτό περιλαμβάνει ρητά και τους ελέγχου των μέτρων που έχουν εισάγει στα εσωτερικά συστήματα ελέγχου τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Και τώρα, εάν προκύψουν οποιαδήποτε ερωτηματικά, υποχρεούμεθα να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όπως αναστολή πληρωμών, διορθώσεις ε, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβιάσεις ε, της ισχύουσας νομοθεσίας. Δεν προτείνουμε βέβαια να υποκαταστήσουμε εμεί τι εθνικέ αρχέ σε καμία περίπτωση. Ταυτόχρονα όμω ορίζουμε σαφώ τι ευθύνε που αναλαμβάνει και η ίδια η Επιτροπή. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, διότι όπως είπα πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ αυτός ο κανονισμός και όσον αφορά τα διοικητικά, τις διοικητικές ακόμα δεν ισχύει, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή τη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση σε ε, επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο ενωσιακό. Τι κάνουμε λοιπόν παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στις εθνικές αρχές και αρρωγή ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι διαχειριστικές αρχές γνωρίζουν απόλυτα όλες αυτές τις ευθύνες όπως ορίζονται. Έχουν προγραμματιστεί για αυτό το σκοπό συναντήσεις στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζουμε στα κράτη-μέλη την υποχρέωσή τους να διαπιστώνουν κατά πόσο τα υπάρχοντα συστήματα έχουν σχεδιαστεί επαρκώς για την ανάληψη τέτοιων ευθυνών και αν αυτό δεν συμβαίνει θα να μεριμνούν ώστε να προσαρμοστούν. Δεύτερον, θα έλεγα ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί οι συγκεκριμένες υποθέσεις που έχουν περιέλθει ε, στη γνώση μας ε, στο πλαίσιο του δικού μας ελεκτικού έργου και του έργου των ε, συναδέλφων μας και οποιασδήποτε καταγγελίες θα αξιολογούνται και θα αναλύονται πολύ αυστηρά. Θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε ελέγχους. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Έλεγχοι για σύγκρουση συμφερόντων έχουν γίνει και στο παρελθόν. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα τομέα όπου θα χρειαστεί να επικαιροποιήσουμε τη μεθοδολογία ελέγχου σύμφωνα με το νέο ορισμό ώστε να ε, μας διασφαλίσουν ε, οι εθνικές αρχές ε, ότι είναι αξιόπιστα όλα αυτά που κάνουν και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να σας ενημερώνουμε για τις εξέλιξεις στον τομέα όποτε και όπου είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, χρυδό χάλια λοιπόν. Δεν με χαροποιεί ιδιαίτερο αυτή η συζήτηση. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα και δεν το έχουμε προσεγγίσει ακόμα. Δηλαδή, είναι το εξή. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν πολιτικοί που έχουν εταιρείε. Ή ένα συγγενή του έχει μια εταιρεία. Και στη μία περίπτωση έχουμε έναν ε, συγγενή ο οποίος ε, έχει πρόσβαση σε κοινοτική χρηματοδότηση. Ε, λέτε 11 με 13 Δεκεμβρίου υπάρχει μια συνεδρίαση, ναι, θα το στηρίξουμε. Βεβαίω το θέμα είναι να πούμε ότι υπάρχουν αυτά τα συστήματα τα οποία βασίζονται ακριβώς στο ότι κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την σύγκρουση συμφερόντων. Τι κάνουν λοιπόν σε όλες τις ε, μέχρι τώρα γνωστές ε, περιπτώσεις ε, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί βεβαίως δεν θα είχαμε περάσει τις ανάλογες διατάξεις. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να εκμεταλλευτούν ευρωπαϊκά κονδύλια στις ε, διαδικασίες ε, των δημόσιων διαγωνισμών, οι οποίοι ήταν στημένοι για να πω το ελάχιστο. Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι τυχαία μέρος σε μια διαδικασία, αλλά για κάτι το οποίο συμβαίνει έσκεμενα. Και ακριβώς για να μην λέμε συνέχεια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, υπάρχει το θέμα αυτό, η υπερόβλεψη αυτή, για να μην λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί αλλιώς θα την εκμεταλλεύονται ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τη θεωρούν ως ε, κάτι το οποίο, ε, απλά, από το οποίο απλά μπορούν να παίρνουν όσα λεφτά θέλουν. Αλλά πάντα βεβαίως αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή η υπόθεση αυτή από τις 11 μέχρι 13 ε, Δεκεμβρίου, εντάξει είναι ευχάριστη, αλλά το καλύτερο θα ήταν να δράσετε αμέσως. αμέσως. Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Το θέμα αυτό το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και δεν θα ήθελα οποιοδήποτε εδώ να έχει την εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει το θέμα ε, με πολύ δραστήριο τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να κλειδώσουν μέσα ε, στα εθνικά συστήματα ελέγχου γιατί εκεί βασίζεται ε, η πρώτη γραμμή άμυνας ε, των οικονομικών κανονισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν θα πρέπει να αξιολογείται και αυτή που χρειάζεται να ενισχύεται. Αυτό πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε ε, πολύ εντατικά με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε πως κάνουν αυτό που χρειάζεται και το κάνουμε. Δεύτερον, και αυτό είναι πολύ πρόημο ακόμα, αλλά σίγουρα χρειάζεται να ελέγχουμε εάν γίνεται επαρκώς και γι' αυτό μας έχει δοθεί η αρμοδιότητα και είμαστε αποφασιστικοί στο να κάνουμε ελέγχους έτσι ώστε τα συστήματα αυτά να έχουν σχεδιαστεί επαρκώς. Και βέβαια βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου αυτή η έλεγχοι και θα γίνουν και για τούτο το θέμα, απερίφραστα. Τώρα είπατε πως υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες υποθέσεις που έχετε στο μυαλό σας και πολλοί που γνωρίζουν τα θέματα αυτά γιατί διαβάζουν τις εφημερίδες και έχουν κάνει θόρυβο. Σε αυτές τις υποθέσεις ε, στεκόμαστε με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπάρχουν μια συγκεκριμένη υπόθεση, για να μην το κρύβω, την οποία σίγουρα έχετε εσείς υπόψη σας που είναι ένας ε, μεγάλος πολιτικός ε, σε κάποιο κρατός έχει καταγγελθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αναλύουμε, το αξιολογούμε με πολύ ενεργό τρόπο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως γνωρίζετε καταρχήν συλλέγει πληροφορίες για όλες τις συμβάσεις που ανατέθηκαν στο συγκεκριμένο όμιλο μέσα στον οποίο έχει οικονομικά συμφέροντα το άτομο αυτό έχει γίνει δύο φορές και τώρα έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τις αναθέσεις, τις αξιολογούμε για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία ότι έγινε κάτι μη σύνομο στα πλαίσια αυτών των αναθέσεων. Για να δούμε τι δράση χρειάζεται. Όποτε ενημερώνεται για κάτι τέτοιο η Κομισιόν, είτε μέσω των media είτε μέσω καταγγελιών, λαμβάνουμε δράση. Χρειαζόμαστε όμως και εμπειρία και στοιχεία για να γνωρίζουμε ότι τα θέματα αυτά βασίζονται όχι σε κάποιες υπόνοιες ή ε, αστοιχείωτες καταγγελίες, αλλά σε πραγματικά δεδομένα. Και αυτό χρειάζεται χρόνο. τον οποίο εμείς διαθέτουμε και θα ήθελα να σας εξασφαλίσω ότι λαμβάνομαι αυτή την ε, ευθύνη πολύ σοβαρά υπόψη. Αλλά δεν βιαζόμαστε να συμπεράνουμε, χρειαζόμαστε να αναλύουμε και να ε, συλλέγουμε πληροφορίε πριν συμβεί οτιδήποτε. Και πότε θα γίνουν οι αναλύσεις. Πότε θα ολοκληρωθούν. Κοιτάξτε. Για την καταγγελία αυτή Ξέρετε πως οι προθεσμίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Μέσα Ιανουαρίου θα πρέπει να επανέλθουμε. Δράση τις επόμενες εβδομάδες λοιπόν. Μόλις έχουμε καταλήξει κάποιο συμπέρασμα. Σας ε, ρωτήσω οι αναλύσεις αυτές ε, τις οποίες λέτε ε, είναι Μιλάμε για την ε, τωρινή καταγγελία, έτσι αυτό είναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριο Στάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση αυτή, το PowerPoint αυτό ήταν ξεκάθαρο και εξηγείται πολύ καλά την κατάσταση για το πώς έχουν τα πράγματα και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η δεύτερη διαφάνεια αφορά την κατάσταση πριν από την Δευτέρα Αυγούστου 2018 και εκεί πέρα λέτε ότι υπήρχε και ο δημοσιονομικός κανονισμός ο οποίος ε, δεν είχε κάποια ρητή διάταξη αλλά υπήρχε μια σειρά πρακτικών ε, που ρύθμιζε σαφώς ε, τα ζητήματα αυτά. Η πρώτη μου ερώτηση είναι λοιπόν ε, η εξής. Στο παλιό κανονισμό είχατε μία ανάλυση ανά κράτος μέλος για το ποιο κράτος μέλος έκανε τι ακριβώς για να προλάβει και να αντιμετωπίσει τις ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Έχετε μία γενική εικόνα στον ε, νέο κανονισμό από ό,τι αντιλαμβάνομαι ακόμα αναλύεται τις ε, πληροφορίες ε, των κρατών μελών. Οπότε η δεύτερη μου ερώτηση είναι η εξής. θα υπάρξει και εδώ πέρα μια ανάλυση ανά κράτος μέλος και η ανάλυση αυτή θα δημοσιοποιηθεί έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης και δημοσιογράφος και βουλευτής θα μπορεί να δει ε, τι γίνεται στο δικό του κράτος μέλος και στα άλλα κράτη-μέλη και ποια μέτρα λαμβάνονται ακριβώς για να προληφθούν οι σύγκρουσεις αυτές συμφέροντων. Αυτή είναι η δεύτερη μου ερώτηση. Η τρίτη μου ερώτηση είναι κάπως πιο συγκεκριμένη και ρητή. Αφορά την περίπτωση ε, για την οποία μιλάμε και τον πολιτικό ο οποίος έχει μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ως εκ της θέσεώς του πρώτος μεταξύ ίσων στην ε, κυβέρνησή του και ήταν ταυτόχρονα ο τελικός δικαιούχος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Στον παλιό ή στον νέο κανονισμό αυτή την στιγμή αυτή τη στιγμή ένας υπουργός ε, πρέπει να εφαρμόζει σωστά τους ε, κανόνες και γίνεται μια καταγγελία θα έπρεπε αυτομάτως να εξετάζουμε υπάρχει εδώ πέρα σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Τώρα ο παλιός ή ο νέος κανονισμός δεν έχει καμιά σημασία. Αν είσαι πρώτος υπουργός, ε, πρωθυπουργός μιας ε, κυβέρνησης τότε βεβαίως ε, το θέμα γίνεται κατεπήγον. Δηλαδή η Κομισιόν θα έπρεπε αυτομάτως να κινείται. Κάνατε κάτι τέτοιο. Τώρα γνωρίζουμε ότι έχει υπάρξει και μια καταγγελία από ανθρώπους από το εν λόγω κράτος μέλος. Τι κάνετε σε αυτήν την περίπτωση. Έχουμε διάφορες γενικές διευθύνσεις οι οποίες είναι αρμόδιες υπάρξει μια συντονισμένη, υπάρχει μια συντονισμένη αντιμετώπιση αυτής της καταγγελίας ή κάθε γενική διεύθυνση που πιθανώς εμπλέκεται η γεωργία και τα λοιπά, περιφερειακή πολιτική, κάνει κάθε μία τα δικά της. Και το ερώτημά μου είναι, υπάρχει κάπου ε, ένα σημείο συντονισμού μεταξύ των ε, γενικών ε, διευθύνσεων. Με άλλα λόγια δηλαδή. Υπάρχει ένας στην Κομισιόν ένα σημείο που τα συγκεντρώνει όλα και αν ναι, ποιος είναι ο υπεύθυνο, ο ένας υπεύθυνο εντός της Κομισιόν και σε διοικητικό επίπεδο, σε ποια γενική διεύθυνση, στη γενική γραμματεία κτλ. Και ο τελικά υπεύθυνο ε, νομίζω είναι ο Επίτροπος Καταπολέμησης της ε, Απάτης, ο κύριος ε, Έτιγκερ. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μου ερώτηση και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση γιατί πραγματικά μας διαφώτισε. Σας ευχαριστώ. πολύ. Είναι πολύ καλές οι ερωτήσεις σας και πολύ σχετικές και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Ξέρετε κι εσείς πως κάνουμε ελέγχους των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και στα πλαίσια του παλιού οικονομικού κανονισμού ήδη τα ελεγκτικά αυτά συστήματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν το θέμα της σύγκρουσης συμφορώντων. Οπότε οι έλεγχοι αυτοί κάλυπταν και αυτή τη διάσταση, όχι όμως αποκλειστικά. Αν είναι απερίφραστα ε, προσβάσιμο και δημόσιο το Μητρό των συστημάτων που έχουν στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω. Θα το σας ενημερώσω μόλις ε, ενημερωθώ κι εγώ. Δεύτερον, θα το εξετάσουμε στο μέλλον, στα πλαίσια του νέου οικονομικού κανονισμού. Όπως σας είπανε, το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, δηλαδή θα συνεργαστούμε πρώτο βήμα με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε πως όλοι έχουν την ίδια ερμηνεία των προτύπων που χρειάζονται και πως τα κράτη-μέλη αυτά ε, τι θα γίνει με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Τώρα, αποτελέσματα ελέγχων. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή η επισκόπηση να είναι δημοσιοποιήσιμη, αλλά πρέπει να επανέλθω στο θέμα αυτό για να δούμε πώς σε επιχειρησιακό επίπεδο θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Η τρίτη σας ερώτηση για το τι θα κάνει σε τρει περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ήδη φαινόταν κάποια σημεία ε, ανησυχίας όπως προσπάθησα να σας πω εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε αναλάβει δράση και έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη που έχουν τις πληροφορίες αυτές να μας στείλουν κάθε μία σύμβαση για τις εταιρείε όπου το άτομο αυτό έχει οικονομικά συμφέροντα. Οπότε ναι, το εξετάζουμε. Για να δούμε σε πρακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο εάν υπάρχουν ε, οποιαδήποτε στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σε ενδεχομένως επόμενα βήματα αλλά δεν θέλω να το προδικάσω γιατί είναι κρίσεις που τρέχουν, είναι ε, συμβάσεις πάρα πολλές τις οποίες ελέγχουμε κάθε μία με λεπτομέρεια και δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Πάντως να είστε σίγουρος πως όπου υπάρχουν τέτοιου είδους σημάδια ανησυχίας ε, θα το κοιτάξουμε γιατί εμείς ως θεσμός έχουμε ευθύνε εδώ. Δεν πρόκειται να τις ε, αφήσουμε στην άκρη. Συντονισμό. Με ρωτήσατε, κάνει ο καθένα τα δικά του ή συντονιζόμαστε. Όχι, συντονιζόμαστε με πολύ προσοχή. Και οι εταιρείε που είναι εδώ συνεργάστηκαν και εγώ με τους συναδέλφους συνεργάζομαι. Έχουμε κάνει και κάποιες συναντήσεις ε, συντονιστικές με τους συναδέλφους για να αντιμετωπίζουμε με διαστρωμένο και συστηματικό τρόπο τα θέματα. Οπότε προφανώς η Γενική Διεύθυνση Budget είναι υπεύθυνη για να εξασφαλίζει πως ο, δημοσιο... ο οικονομικός κανονισμός εφαρμόζεται σωστά, αλλά επίσης έχουμε μέτρα τα οποία έχουν λάβει μεμονωμένες, που έχουμε λάβει για μεμονωμένες αποφάσεις που για ε, κάποιον ε, υπόλογο στην Κομισιόν έχουν ε, ληφθεί αποφάσεις και αυτό βέβαια έχει να κάνει με κάθε γενική διεύθυνση που είναι αρμόδια. Και γι' αυτό είναι ο συντονισμό τόσο σημαντικό. Άλλωστε. Και γι' αυτό τον παίρνουμε τόσο στα σοβαρά. Το οποίο σημαίνει ότι σε επίπεδο πολιτική ευθύνη οι δικέ μα ε, οι αρχικά μας ε, ε, ανώτεροι έχουν τις δικές τους ευθύνες. Ο κύριος Έτενκερ, για παράδειγμα, είναι αρμόδιος και για τα θέματα διερμηνίας και για τα θέματα απάτης και για τον οικονομικό κανονισμό, ενώ υπάρχουν και άλλοι ε, επίτροποι που είναι για τις επιχειρηγήσεις και τις επιδοτήσεις που δίνονται στο δικό του τομέα στα επιχειρησιακά θέματα αρμόδιοι. Οπότε και αυτοί θα πρέπει να συναντηθούν για να τα παρακολουθούμε όλα στενά και να ξέρουμε πως η απόκριση που δίνουμε ε, εγκάρσια είναι η σωστή. Ωραία, θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο το ιστορικό. Το 2014 σε μια επίσκεψη στη Τσεχική Δημοκρατία υπήρχε ένας υπουργός Οικονομικών ο οποίο ήταν ο ίδιο ένα μεγάλο δικαιούχο και για μένα ω Γερμανίδα, αυτό ήταν αδιανόητο. Έχουμε σχετικό η νομοθεσία στη Γερμανία που απαγορεύει κάτι τέτοιο. Είναι αδιανόητο σε ένα κράτο μέλο ε, να επιτρέπεται κάτι τέτοιο για μένα. Τότε λοιπόν στην επίσκεψη στην Τσεχία διαπραγματευτήκαμε και μιλήσαμε με την ελεγκτική αρχή. Και όταν φύγαμε, άλλαξε η ελεγκτική αρχή. Όχι μία φορά, πολλές φορές. Και όταν πήγαμε να ψάξουμε να βρούμε ποιο ήταν το πρόβλημα, τότε μάθαμε ότι είχαν υπάρξει παρεμβάσεις πολιτικές από τον πολιτικό δικαιούχο στις ελεκτικέ εργασίες. Έτσι μάθαμε τότε. Μετά, σε αυτό το κράτος μέλος, ε, ο τύπος είναι πολύ δραστήριος και ο τύπος λοιπόν ανέφερε τους, ε, τους έβαλε μια παγίδα ουσιαστικά. Και κατάφερε να ανακαλύψει ποιος ήταν ο πραγματικός δικαιούχος, ο επιχειρηματίας δηλαδή, και ότι υπήρχε παραβίαση της Ευρωπαϊκής Δομοθεσίας. Οι μέτοχοι ήταν τα παιδιά του και ε, αυτή η ποινική διαδικασία λοιπόν πήρε την πορεία της. στην Κρυμαία λοιπόν. Και πίστηκε τότε το κοινοβούλιο ότι υπήρχε ασυμφωνία μεταξύ πολιτικών και επιχειρήσεων τέτοιων και επιχειρηματιών όταν δρούν ως πολιτικοί. Στην Τσεχία το έκαναν λοιπόν μετά από σκληρές ε, εργασίες, σκληρές προσπάθειες. Πίστηκε η κυβέρνηση της Τσεχίας να το υλοποιήσει αυτό, να μην υπάρχει δηλαδή μόνο στο χαρτί. Είχαμε άρση ασυλίας με δραματικές εξελίξεις ε, και εμένα πάντα μου κάνει έκπληξη όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Μετά κατέστησε αφές ότι η υπόθεση αυτή υπήρξε και έρευνα της Όλαφ έμεινε ατιμόρυτη παρά τα στοιχεία απάτης. Μέχρι και σήμερα με συγκλονίζει το ότι ήταν σημαντικό το ποινικό αδίκημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Η Γενική Διεύθυνση Ρέτζη ε, ε, συζήτησε και με τον Επίτροπο και τώρα που είμαστε σήμερα, σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ο ίδιος δικαιούχος που κανονικά είχε τεθεί σε μαύρη λίστα για πολλά χρόνια, εξακολουθεί να λαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αυτό προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά πρέπει να πω ότι οι δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν τότε με αυτή την υπόθεση μιλήσαμε εκεί πέρα και με τους ε, ελεγκτές, ε, λάβαμε τα email και δεν είδαμε να υπάρχει κάποια ανάληψη της ευθύνη από τον πολιτικό. Αυτά τα πράγματα ήταν ήδη γνωστά. Δηλαδή τι πρέπει να συμβεί για να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι όροι, όροι οι οποίοι ε, παραβιάζονται εδώ και χρόνια. Δηλαδή παριστάνουμε τους ηλίθιους σαν να μπορούμε να πούμε ε, ότι 2 και δύο κάνει 4. Πραγματικά σοκάρομαι και η άλλη περίπτωση με τον ε, γαμπρό, ε, τον συγγενή δηλαδή. Είναι τα πράγματα, είναι προφανή και μιλάνε από μόνα τους. Γνωρίζετε Εντάξει, τι είναι σημασία των κρατών μελών. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ναι, το ελέγξαμε και τα λοιπά. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, Πού θα πάει αυτή η υπόθεση. Ανησυχώ γιατί το γεγονός ότι έχουν φτάσει τα πράγματα ως εκεί ε, είναι και ζήτημα δικαιοσύνη στη συγκεκριμένη χώρα. Σε άλλες ε, χώρες ε, δεν θα φτάναν ως εκεί να βάζει κάποιος το, το χέρι στο μέλι τόσο απροκάλυπτα. δεν είναι δυνατόν δηλαδή να Εντάξει, εκκλήσει και τα λοιπά, ξέρω ότι δεν καταφέρνουμε τίποτα έτσι, αλλά ξέρουμε προ τα πουν ε, πάνε τα πράγματα και αυτή η, η αμηχανία της ε, Κομισιόν ε, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο με απογοητεύει. Γιατί εδώ πέρα αποτυγχάνουμε σε μια σε ένα γενικότερο φαινόμενο που κάποιοι άνθρωποι απλά παίρνουν τα ε, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βάζουν στην τσέπη και πλουτίζουν. Θέλετε να πείτε κάτι. Κοιτάξτε, συμφωνώ με τις ανησυχίες σας ότι κάτι πρέπει να γίνει και να το δούμε σοβαρά. Όπως είπα, Δηλαδή αν δούμε το τι γινόταν στο παρελθόν είναι σαφές ότι το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Ε, θέλω να είμαι σαφής. Το εξετάζουμε αυτό όπως σας είπα από κοινού. Εξελογούμε όλες τις συμβάσεις ε, και επί της βάσης αυτής ε, δεν θα απαιτηθούμε των ευθυνών μας και δεδομένου του ότι όλες αυτές οι κατηγορίες αφορούν διατάξεις ε, με το παλιό καθεστώς αλλά και με το παλιό καθεστώς παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες απαιτήσει ε, για τα συγκρόμενα συμφέροντα όμως πρέπει να είμαστε σαφείς παρά το ότι πράγματι η εικόνα που δίνεται είναι άθλια το κριτήριο τελικά είναι το εάν νομικά έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία επαρκούν για να αναλάβουμε δράση. Σε τελική ανάλυση είμαστε υπό το κράτος δικαίου και αυτό είναι κάτι το θετικό. Πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε πάρα πολύ υψηλέ προδιαγραφές στην αξιολόγησή μας αυτή και όπως είπα αυτό ακριβώς κάνουμε μέσω αυτής της κοινή επιχείρησης των αξιολογήσεων αυτών δεν νομίζω ότι συμβαίνει επί μου βάσεως ε, να συλλέγουμε στοιχεία για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν μια συγκεκριμένη επιχείρηση και να τις αναλύουμε μία προς μία κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα προφανώς η έκθεση την οποία αναφέρατε Ναι, Βεβαίω είναι ενισχυτικά αυτά τα οποία προκύπτουν για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια νομική ανάλυση και θα γίνει στο πλαίσιο της ε, ανάλυσης που κάνουμε τώρα. Για το μέλλον, ε, μιλήσατε ακριβώς για προφανείς ε, δυσκολίες. Ε, το δεν θέλω να επισέλθω σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά μιλώντας, όταν τα μέλη μια κυβέρνησης, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, βλέπονται σε καταστάσεις όπου λαμβάνονται οικονομικές αποφάσεις που μπορούν να τα ωφελήσουν αμέσως ή εμέσως, τότε ακριβώς ο δημοσιονομικός κανονισμός απαιτεί να λάβουν δράση για να διορθωθεί αυτό. θα πρέπει ακριβώς ε, να προσέχουμε να μην ε, συγχαίουμε καταστάσεις ε, όπου ίσως έχουμε περιπτώσεις αντικρώμενων συμφερόντων. Ε, που δημιουργούν νομικές δυσκολίες με άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα πράγματι αποτελεσματικής ε, αντιμετώπισης. Ε, μία τέτοια αποτελεσματική αντιμετώπιση θα μπορούσε να είναι παραδείγματος χάρη ένα καταπίστευμα το οποίο θα έχει δημιουργηθεί κατά τρόπον ώστε ο λόγο λόγω δεν θα ξέρει το τι περιέχει και ποιες αποφάσεις λαμβάνονται από αυτό. Σε τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, δεν μπορεί πλέον να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ε, πάρμιος και ανάλογα και με το εθνικό νομικό σύστημα μπορούν να απέχουν πλήρως η πολιτική από την λήψη αποφάσεων και αυτό γίνεται σε κάποια κράτη-μέλη. Ακριβώς ε, λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε εάν ε, αυτά τα οποία προσφέρονται ως τρόποι αντιμετώπισης ανταποκρίνονται σε αυτές τις υψηλές προδιαγραφές και έχουμε τώρα και τα νέα άρθρα του Δημοσιονομικού Οργανισμού που είναι πολύ πιο λεπτομερή και συγκεκριμένα και κάνουν και πιο εύκολη τη δουλειά μας. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μιλήσατε για το μέλλον. Το παρελθόν έχει κλείσει, τα χρήματα πέταξαν. Ξεκινώντας από το παράδειγμα που έδωσε η κυρία Γκρέτσλερ για αυτόν τον Υπουργό προϋπολογισμού που έκανε ό,τι έκανε, θα έλεγα ότι δεν πρόκειται εδώ για παρόμοια περίπτωση. Ουγγαρία, Ρουμανία. Αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες και το γνωρίζετε. Έχει χρόνια που συμβαίνει και συμβαίνει ακόμα. Επίση, ψάξτε αυτούς που δεν έχουν τα χρήματα αυτά σε επιχειρήσεις στο όνομά τους, αλλά επιχειρήσεις με ονόματα τρίτων, παρόλο που αυτοί λαμβάνουν τα χρήματα. Γιατί αν ο κανονισμός λέει δεν έχετε δικαίωμα ε, να λάβετε χρήματα αν είστε πολιτικός, ε, θα βρεθεί κάποιος να σας καλύψει. Αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να κακοδιαχειριστούν τα ευρωπαϊκά ταμεία θα βρούνε τρόπους. Το αίτημα της αποχής ε, με ιδία δήλωση μπορεί σε κάποια ένα-δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί αλλά στα άλλα όχι. Τι, ε, θα πω εγώ ότι απέχω τη στιγμή που έχω σκοπό να κλέψω, θα το κάνω με άλλο τρόπο, γιατί έχω την εξουσία. Και μην ξεχνάτε πως η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία και στη Βουλή συνήθως, οπότε δεν πρόκειται να ψηφίσει τέτοιου είδους νομοθεσία. What I would say is... Αυτό που θα έλεγα στην περίπτωση αυτή είναι πως το νομικό πρότυπο θα πρέπει να είναι να υπάρχει αποτελεσματική ε, ε, δράση ε, αποκατάστασης. Αυτό. Τώρα, συγκεκριμένες υποθέσεις είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κανονισμός και θα έχει τα δικά του διορθωτικά μέτρα και θα έχει άμεση εφαρμογή στα κράτη-μέλη με υποχρέωση αποτελεσμάτων. Τώρα, τι είναι αποτελεσματικό διορθωτικό μέτρο ένδικο μέσο σε συγκεκριμένη χώρα, σε συγκεκριμένο κράτο μέλο, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί σε άλλη περίπτωση να μην είναι διορθωτικό, ναι, ε, αποτελεσματικό. Αλλά η απέτηση να παράσχουμε αποτέλεσμα παραμένει. Και αυτό είναι το πρότυπο επί του οποίου θα κρίνονται αυτέ οι υποθέσει. Καταγράφω αυτό που λέγεται, είναι πάρα πολλέ οι δυσκολίε όντω σε πολλά κράτη-μέλη. Με του πολιτικού και τα χρήματα, προφανώ δεν μπορώ να το σχολιάσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως οι νέοι κανόνες στο σημείο αυτό και εσείς παίξατε πολύ μεγάλο ρόλο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον οικονομικό κανονισμό όταν εγκρίθηκε αυτός. Είναι σημαντικό, είναι ε, πολλές οι απαιτήσει που προκύπτουν και είναι εφαρμοστέο άμεσα από τα κράτη-μέλη. Και εμάς η υποχρέωσή μας είναι να εξασφαλίσουμε πως τα ευρωπαϊκά χρήματα ε, προστατεύονται με αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των κανόνων. Και αυτό έχουμε στόχο να κάνουμε στο μέλλον. Σα υπενθυμίσω ότι ναι, αυτό το οποίο είπατε για ένα τυφλό καταπίστευμα νομίζω μας έδωσαν μια διαβεβαίωση σχετική το 15-16 και λέμε εντάξει έληξε. Αλλά μετά μάθαμε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονταν από το ίδιο άτομο πάλι. Ε, πρέπει να ρυθμιστεί αυτή η υπόθεση θα πρέπει η Κομισιόν να αναλάβει τις ευθύνες της. Αυτή είναι η βούλησή μας και συνοψίζοντας την συζήτηση, η συζήτηση αυτή δεν έχει τελειώσει και είμαστε αποφασισμένοι να γίνει αυτή η συζήτηση γιατί είμαστε πεπισμένοι πως εδώ πέρα παίζεται αυτό το οποίο αποκαλούμε πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε άτομα τα οποία παραβιάζουν ανοιχτά τους ε, κανόνες. Ε, βλέπουμε ότι έχουμε δεσμούς ξεκάθαρους με τις εταιρείε από άτομα σε ηγετικές θέσεις που προσπαθούν μετά να επηρεάσουν ε, και την περιφερειακή πολιτική. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής ο Αρμόδιος εκεί πέρα Ήδη λοιπόν αφήνει μια πολύ πικρή γεύση η όλη αυτή η υπόθεση. Θα πρέπει ε, να δούμε αυτό το θέμα κατεπηγόντως και θα το παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά και οπωσδήποτε μέχρι τον Ιανουάριο που θα τα ξαναπούμε αναμένουμε κάποιες ε, εξελίξεις. Και αναμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνές σας. ευχαριστώ όλους ε, που ήρθατε. Ήσασταν τυχεροί, τα ανέλαβε όλα ένας ε, συναδελφός σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Θα έρθουμε το απόγευμα με την ακρόαση του κύριου Σέλμαϊρ.